La récréation est terminée. Τέλος το διάλειμμα. Mesdames, Messieurs. Κυρίες και κύριοι, κυρίσω την έναρξη συνεδρίασης. Είμαστε απευθείας στο διαδίκτυο και όλος ο κόσμος έχει το βλέμμα του στραμμένο επάνω μας. Ιδιαιτέρως στο Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλωσορίζω τους εκπροσώπους τους. Λοιπόν, Σήμερα το πρωί έχουμε πάρα πολύ σημαντική συνεδρίαση, διότι θα κληθούμε να εγκρίνουμε τις τροπολογίες σε δεύτερη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ για την πολυπληθή σας παρουσία. Θα μπορούσαμε να είμαστε και περισσότερο, δεν πειράζει. Μπας Μόλις τελειώσουν το πρωινό τους, θα έρθουν και άλλοι συνάδελφοι. Euh, σας ζητώ πρώτα απ' όλα να δώσετε πολύ μεγάλη προσοχή διότι θα σας εξηγήσω τα έγγραφα επί των οποίων θα εργαστούμε και στη συνέχεια θα ήθελα επίσης να σας παρακαλέσω να προετοιμαστείτε ψυχολογικά για να ψηφίσετε πράγματα που δεν θα καταλαβαίνετε. Είμαστε σε ένα δημοκρατικό σύστημα και διαφανές θυμίζω. Αλλά τα ε, δημοσιονικά προβλήματα δεν είναι περίπλοκα, είναι βιβλικής απλότητας. Παίρνουμε από ε, το ένα κονδύλι για να δώσουμε στο άλλο. Σε αυτό ανάγεται όλη η υπόθεση. Αλλά για να γίνει αυτό, ο μηχανισμός είναι περίπλοκος. Και είναι πολύ περισσότερο περίπλοκος που έχουμε εκατοντάδες γραμμές στον προϋπολογισμό και χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στην ειδική πλειοψηφία στην Ολομέλεια και ακόμα καλύτερα στη ευρύτερη δυνατή πολιτική συνένεση χρειαζόμαστε λοιπόν την εξασφάλιση ότι κάθε ομάδα θα επιτύχει αυτό που την ενδιαφέρει περισσότερο στα πλαίσια του συμβιβασμού και της συνένεσης. Βεβαίως, θα πρέπει να βεβαιωνόμαστε πάντα ότι οι ε, πολιτικές προσαρμογές της τελευταίας στιγμής που κάναμε χτες το βράδυ στους συντονιστές είναι πλήρως συμβατές με την ε, συμφωνία της ιδιαλλαγής και τη σέβονται και δεν την παραβιάζουν. Συμφωνία ε, με το Συμβούλιο. Λοιπόν, είναι περίπλοκη η παρουσίαση, συνεπώς και εγώ μπορώ να σας διαβεβαίωσω ε, πάση περιπτώσει ότι μαζί με τους συντονιστές και όλους μας τους συνεργάτες και ευχαριστώ και τη γραμματεία και τους υπαλλήλους των πολιτικών ομάδων εργαστήκαμε με τρόπο ώστε όλα αυτά να γίνουν ε, με πλήρη διαφάνεια, πλήρη κατανόηση από όλου. Και αν υπάρξει κανένα σφάλμα που έχει πάρει σπίση, θα είναι τεχνικό. Μόλι ε, ρυθμίσαμε ένα με το Συμβούλιο. Ξέρετε ότι η οι υπολογιστέ δεν βγάζαν τα ίδια αποτελέσματα. Το Συμβούλιο έλεγε 2 και 2 ίσον 5, οι δικοί μα υπολογιστέ έλεγαν 2 και 2 ίσον 4 και βρήκαμε το σωστό υπολογιστή. Présentation des documents. Πρώτον, παρουσίαση των ε, εγγράφων που ε, λάβατε χτες, που φυλάξατε με μεγάλη προσοχή, το βάλατε στο μαξιλάρι σας και κοιμηθήκατε για να μην σας το πάρει κανένα στο έγγραφο αυτό και μετά φέρατε το φάκελο μαζί σας. Είναι το λεγόμενο έγγραφο υπαριθμών 9. για την ψηφοφορία στη δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου. Σήμερα το πρωί αυτό το έγγραφο μας είναι τελείως άχρηστο. Μπορείτε να καθίσετε πάνω του. Πάντα με μεγάλο σεβασμό τον οποίο οφείλουμε στο Συμβούλιο. Αλλά δεν θα το ψηφίσουμε αυτό το έγγραφο. Υποκλεινόμαστε με σεβασμό. Κοιτάξτε το και δεν θα το ξαναδείτε ποτέ. Ξεχάστε το μετά για πάντα. Είναι το δεύτερο, η δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου και το βάζουμε σε αρχείο. Είναι γραφείο αναφορά. Βάλτε τη σιγαρέκλα, καθίστε πάνω του και ξεχάστε το. Δεν θα το ξανασυζητήσουμε. Άλλο θέμα. Πολύ πιο σημαντικό τώρα το έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να ψηφίσουμε. Είναι το υπαριθμό 10. Είναι αυτό το παραλληλεπίπεδο, το γόνιο παραλληλεπίπεδο. Ε, η μία του πλευρά είναι μεγαλύτερη από την άλλη. Και τρία παραρτήματα, ένα, δύο και τρία, του εγγράφου υπαριθμών 10 έχει αυτή τη μορφή που σας δείχνω, επαναλαμβάνω ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, δεν είναι τετράγωνο και είναι ο κατάλογος όλων των τροπολογιών στο έγγραφο υπαριθμών 10. Μην το πετάξετε αμέσω. θα το χρειαστούμε ίσως. Και αυτό το έγγραφο λοιπόν υπαριθμών 10 είναι Ε, όλες μας οι τροπολογίες της πρώτης ανάγνωσης που θα τις χρειαστούμε. Είναι λοιπόν ε, οι πίνακες και τα βαρτήματα. Το σημαντικότερο όμως έγγραφο δεν το είδατε ακόμα. Που είναι η τροπολογία στη δεύτερη ανάγνωση που επίσης επιγράφεται 10, αλλά 10 ραπ. Ραπ όπως λέμε ραπορτέρ, δηλαδή εισηγητής. Και τα αντίστοιχα τετράδια, τετράδια, ένα έγγραφο είναι. Λοιπόν, έχετε το πίνακα που λέει τροπολογίες δεύτερης ανάγνωσης του εισηγητού 10 ραπ και τις λεπτομέρειες που είναι επίσης 10 ραπ αλλά είναι το παράρτημα στο προηγούμενο και ένα τελευταίο τώρα. Ένα τελευταίο λέγω. Έχουμε ένα φύλλο, ένα πίνακα, ένα σκέτο χαρτί. Πρώτη Δεκεμβρίου, 20 ώρα και τέταρτο λέει εδώ. Και αυτό τι είναι? Τροποποίηση τελευταία στιγμής στο 10 και στο 10 ραπ. Είναι τα πρακτικά συμπεράσματα και τα συγκεκριμένα της πολιτικής ολοκλήρωση και συμπεράσματος στο οποίο χτες καταλήξαμε με τους συντονιστές. Εντάξει, αυτά λοιπόν είναι τα έγγραφα και θα αρχίσουμε στη συνέχεια με την εξέταση των προφορικών τροπολογιών γιατί έτσι χαρακτηρίζονται αυτά νομικά, προφορικές τροπολογίες του εισηγητού, σε σχέση με το έγγραφο 10 και 10 ραπ. Λοιπόν, αρχίζουμε από το ε, φύλλο αυτό, σας προτείνω, και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε πιο εύκολα, Ο ΜΟΥ ε, έγραφα 10 ραπ και 10 σκέτο ε, με την επιφύλαξη κάποιων βεβαίως κατά τμήματων ψηφοφορίων, κατά που μας ζήτησαν οι πολιτικές ομάδες και θα τις ε, δούμε τη μία μετά την άλλη. Ωραία. Για τα έγγραφα, το καταλάβαμε αυτά. Ερωτήσεις έχετε, έχετε όλοι τα έγγραφα στα χέρια σας. Αισθάνεστε όλοι ανετά με τους καταλόγους αυτούς. Εάν ναι, καλώς. Κατά τα άλλα μπορούμε να κατρακυλήσουμε την πλαγιά και να ψηφίζουμε μηχανικά και αυτόματα χωρίς να καταλάβουμε περισσότερα από αυτά που θα μας λέει ο εισηγητής. Και δίνω το λόγο στον εισηγητή μας. Ε, thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ήμουν παρατηρητής εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έψαχνα μία αίθουσα στο Στρασβούργο και ρώτησα κάποιον πού είναι αυτή η αίθουσα. Και μου είπε, μη με ρωτάτε, εγώ δέκα χρόνια είμαι μόνο εδώ. Κάπως έτσι έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ακούγοντας λοιπόν εχθές τους συντονιστές με στόχο να έχουμε όσο δυνατόν ευρύτερη συνένεση, έκανα κάποιες αλλαγές τις οποίες συζητήσαμε μετά που λάβαμε αυτόν τον πίνακα. Αν δεν κάνω λάθος έχουμε 7 σημεία προς διευκρίνηση. Το πρώτο αφορά τη γραμμή 040304 για το EURES. Αυτή είναι τροπολογία Είχαμε συμφωνήσει για τις δεσμεύσεις στον τίτλο 1α. Ζητώ συγγνώμη κύριε Σιγητά. Τα μέλη μπορούν να παρακολουθούν αυτά που λέει μα στον πίνακα αυτό. Et donc, la ligne qui est... Είναι η πρώτη γραμμή λοιπόν με γκρι από πάνω. Θα σας μιλήσει ο εισηγητής για τις αλλαγές μετά τη συμφωνία που έγινε χτες το βράδυ με τους συντονιστές και βλέπετε ότι έχουν υπογραμμιστεί με γκρι και φαίνονται καλύτερα το σε αυτές. Συγγνώμη κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. The message is that in this line... Λοιπόν, το μήνυμα είναι ότι σε αυτή τη γραμμή θα πρέπει να ε, αυξήσουμε την πληρωμή κατά 700 για να έχουμε ε, ταύτιση με τις δεσμεύσεις. Ο κύριος Γκοτμάνης, με συγχωρείτε για να καταλάβω καλά γιατί μιλάτε. Πρέπει να πάρουμε το 10 της δεύτερης ανάγνωσης, γιατί στο 10 AP δεν συμπεριλαμβάνεται αυτό. Και εδώ έχουμε συν 500, όχι με συγχωρείτε, συν 1 εκατομμύριο δεσμεύσεις, συν 700 πληρωμές. Και θα μείνουμε σε αυτό που έχουμε εδώ στον πίνακα. Επιβεβαιώνει ο εισηγητής. So amendment... Αν δείτε λοιπόν την τροπολογία στη γραμμή αυτή, συμφωνήθηκε η δέσμευση για την άλλη γραμμή, αλλά προκειμένου να έχουμε το ίδιο ποσό ή τουλάχιστον ένα λογικό ποσό της πληρωμής, θα πρέπει να το αυξήσουμε. Όπως είπε ο κύριος Γκοντμάνες, στο έγγραφο 10, 10 πρόκειται για τη σελίδα 9. Πρόγραμμα, πρόγραμμα Eures, όπως είπε ο εισηγητής. Θέλουμε πληρωμές υψηλότερες από αυτές τις οποίες είχε προβλέψει το Συμβούλιο. 19 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στις υποχρεώσεις και 16 εκατομμύρια στις πληρωμές, ενώ το Συμβούλιο μιλούσε για 15 εκατομμύρια 300.000 ευρώ σε πληρωμές. Και ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραμείνει αυτή η τροπολογία, να μην αποσυρθεί. Η επόμενη είναι για τις παρατηρήσεις στη γραμμή 070401 για το Δημοσιονομικό Μέσο Πολιτικής Προστασίας. Δεν υπάρχουν ε, δημοσιονομικές επιπτώσει επ' αυτού, αλλά για να έχουμε ό,τι είχαμε και στην πρώτη ανάγνωση θα πρέπει να παραμείνει. Το τρίτο είναι το 140303, ε, τίτλος 4, ως μέλη σε διεθνείς οργανώσεις ε, ε, τελωνιακές και φορολογικές. Αυτή θα πρέπει να παραμείνει και όχι να αποσυρθεί όπως έχουμε στην αρχικό πίνακα. Η τέταρτη είναι η 150203. Εδώ είναι μια τεχνική διόρθωση, είναι ένα λάθος της μετάφρασης και εδώ συμφωνήσαμε ότι είναι λογικό να τη δεχτούμε. Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα στο οποίο υποστηρίζονται φοιτητές και μαθητές και ε, στην αγγλική εκδοχή υπήρχε ο όρος personal, personnel, συγγνώμη, ε, και δινόταν ίσως η εντύπωση ότι οι εργαζόμενοι στον οργανισμό αυτό έλαμβαναν τα κονδύλια και για να μην δημιουργείται αυτή η σύγχυση επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την τεχνική αλλαγή και κατόπιν λάβαμε μία επιστολή από τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού, από την πρόεδρο, ότι τους ικανοποιεί η εξήγηση για τις ανακοινώσεις. Επομένως, ε, οι επιφυλάξεις ε, για τις δύο ανακοινώσεις που είχαν ανακοινωθεί στην πρώτη ανάγνωση άρονται. Αυτό συμφωνήθηκε και στις συνεδρίες των συντονιστών. Κατόπιν, έχουμε μία γραμμή στις δημοσιονομικές υπηρεσίες 12.04.01 και εδώ υπήρχε ένα μικρό ε, ποσό ως περιθώριο στον τίτλο 1α. Υπήρξε πρόταση από κάποιες ομάδες, ε, τμήμα αυτών των χρημάτων, να πάνε στις δημοσιονομικές υπηρεσίες. Όταν επιστρέψαμε στον αρχικό προπολογισμό στον τίτλο 1α, υπήρχε κάποιο αποθεματικό. Και το προσχέδιο προπολογισμού και αποφασίσαμε να μην το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό το περιθώριο χρησιμοποιήθηκε εν μέρη για τη χρηματοδότηση των μικροπιστωτικών ε, και μας περίσσεψαν και 10 εκατομμύρια. Αυτά τα 10 εκατομμύρια πήγανε στις λεγόμενες γραμμές προτεραιότητες ε, για τις οποίες συμφώνησαν οι συντονιστές και κατόπιν αυτή της κατανομής, η οποία έγινε αναλογικά, ανάλογα με το ε, βάρος αυτών των γραμμών, μας είχαν περισσέψει 706.000 και πρόταση είναι πλέον οι 560 από αυτό να πάνε στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Και έτσι έχουμε επιπλέον 700. Τέλος, για την ΚΕΠΑ είχαμε ε, μία περικοπή κατά 150.000 ευρώ και η περικοπή αυτή δεν συνάδει με τη συμφωνία που είχαμε στην ε, συνδιαλλαγή. Επομένως, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την περικοπή pacta sunt servanda. Δεν υπάρχει πρόβλημα για την ανάληψη υποχρεώσεων, γιατί υπάρχει σχετικό περιθώριο στον τίτλο 4, που σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων και μειώνεται το περιθώριο για τον τίτλο 4. Είναι διαχειρίσιμη αυτή η περικοπή. Υπάρχουν και κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν απαραίτητο ε, στις πληρωμές για κάποιους υπολογισμούς που δεν είναι απολύτως σωστοί. Και μετά από πρόταση και της γραμματείας, ο εισηγητής προτείνει η πληρωμή, οι πληρωμές της γραμμής 081001, που είναι σχετικά μεγάλη γραμμή προϋπολογισμού, 540 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή τη φάση να τη χρησιμοποιήσουμε ως ε, μαξιλαράκι. Και η απαραίτητη μείωση πληρωμών για να επιτύχουμε το συμφωνημένο περίπου 123 δις ε, των πληρωμών σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουμε αυτά τα 540 εκατομμύρια στην 11.009.000 που περιλαμβάνει και την ΚΕΠΑ. Και κατόπιν κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι αν σε αυτή την ε, ψηφοφορία δεχτούμε και τα όσα μας είπε η Επιτροπή Πολιτισμού, μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα και στο ψήφισμα. Υπάρχει ένα σημείο στο ψήφισμα, το οποίο ασχολείται με, το, με τις επιφυλάξεις και όλη αυτή την ιστορία με τις ανακοινώσεις και εκεί ο εισηγητής προτείνει κατά τμήματα ψηφοφορία για να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε και με την πρόσφατη απόφαση. Δεν θέλω να περιπλέξω τα πράγματα περαιτέρω, γι' αυτό λοιπόν προτείνω μετά την ε, ψηφοφορία unblock να ψηφίσουμε κατά τμήματα κάποια σημεία που ήταν αιτήματα συγκεκριμένων ομάδων. Δεν μπορούμε να τις ε, ψηφίσουμε όλες μαζί και αυτές γιατί καταλήξαμε σε αυτή την άποψη. Έχουμε κατά ψηφοφορία γιατί η μία ή άλλη ομάδα έχει διαφορετική άποψη και ε, θα πρέπει να προσπαθήσουν να περάσουν αυτή την άποψη είτε ε, ψηφίζοντας κατά τμήματα είτε βλέποντας τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, θα ζητώ να ψηφίσετε αυτές τις αλλαγές που σας ανέφερα. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Ήταν όντως πολύ σαφή, στο βαθμό του δυνατού τουλάχιστον. Και απόλυτα σύμφωνα με τον πίνακα αυτόν, τον οποίο μας παρουσιάσατε και σχολιάσατε τώρα. Όχι, όχι, όχι, δεν ήταν, παρακαλώ. Σχεδόν, πρόεδρε, σχεδόν, σχεδόν να αρισμονήσω να αναφερθώ στο τεχνικό τμήμα, γιατί αναφέρθηκα στην ουσία της ΚΕΠΑ, αλλά όχι στο τεχνικό. Έχουμε μία γραμμή που δεν είναι γκρίζα, 19.01.04.04. Αυτή αποσύρεται. Αναφέρθηκα ω προ το περιεχόμενο, αλλά όχι με, τον με ποιο τρόπο προτείνω να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Καλώ, λέει ο Πρόεδρο. Επαναλαμβάνω για το Συμβούλιο ότι οι τελευταίες προτινόμενες ε, προσαρμογές εξασφαλίζουν απόλυτα σχεδόν το σεβασμό των αποτελεσμάτων της συνδιαλλαγής με την ε, ΚΕΠΑ σε 281 ε, μισό εκατομμύρια σε αναλήψεις υποχρεώσεων και ο προσδιορισμός του συνολικού ποσού των πιστώσεων πληρωμών για το σύνολο του προπολογισμού ανέρχεται σε 122 δισεκατομμύρια 937 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί ήταν τα προβλήματα των υπολογισμών και των υπολογιστών. Διευθετούνται λοιπόν τα προβλήματα αυτά και κυρίως για να καλυφθεί το συνολικό όριο των 123 δις των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων, στο οποίο συμφωνούμε. Έχουμε την προφορική τροπολογία με το γκρι χρώμα στον πίνακα, στο αριστερό τμήμα, στο αριστερό κάτω τμήμα του πίνακά σας, όπου έχουμε περίπου 4 εκατομμύρια πληρωμές από μια γραμμή με ένα πολύ όμορφο και ελκυστικό όνομα, πρόγραμμα ιδεών. Πρόκειται για την χρηματοδότηση που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στους φωτεινότερους νόες της Ευρώπης, τους καλύτερους επιστήμονες. 536 εκατομμύρια 900.000 ευρώ για αυτό τον ειδικό ε, για αυτήν την ειδική χρηματοδότηση για να παραμείνουν οι ιδέες που θα διαδοθούν και θα αναπτυχθούν στην Ευρώπη στο ύψιστο επίπεδο και για το 2010. Ο κύριος ε, Γκότμαν έχει δει το λόγο. Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Έχω δύο <laughs> ερωτήσεις προς τον συγγητή. στη γραμμή 08-1001. Ποιο είναι το τελικό νούμερο στις πληρωμές. 540 εκατομμύρια μείον 5 εκατομμύρια. Ψηγητής. Αν δεν κάνω λάθος και παρακαλώ να με ελέγξει ο Καρλ, είναι το τελικό νούμερο 536.009.000, δηλαδή 536 εκατομμύρια 9.000 ευρώ. Καλώς, ευχαριστώ πολύ και για τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Γιατί εμεί είχαμε στήσει ένα εκατομμύριο, 100.000 ε, μάλλον επιπλέον στην αρχή. Έχει αλλάξει αυτό από ό,τι φαίνεται με την πολιτική συμφωνία. Το τελικό νούμερο ποιο είναι. Μέχρι χθε ήταν 4,4 εκατομμύρια. Τώρα τι, προσ, τι προστίθεται, 560 Αύξηση έχουμε, λέει ο κύριος ε, Σόριαν. Είμαστε πάνω από το προσχέδιο. Από τα 10 εκατομμύρια που ανέφερα νωρίτερα, διανύμαμε τα 140. Και μαζί με αυτά τα 140 τώρα βρισκόμαστε σε επίπεδο 700 επιπλέον του ε, προσχεδίου. Στις πληρωμές έχω 4.400.000. Καλώς, σαφές το νούμερο, ευχαριστώ. Πρόεδρος, ως εκ τούτου, εάν γίνει η τροπολογία, στην οποία ιδιαίτερα αποδίδουν σημασία οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι συνάδελφοι, και οι φιλελεύθεροι βεβαίως βεβαίως, το συνολικό ποσό στον προπολογισμό σε αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχεται σε 6 εκατομμύρια και στις πληρωμές 4 εκατομμύρια 400.000. Είμαστε εντάξει κύριε Σεγητά. Ναι. Αλλά η ερώτηση θα είναι οι πληρωμές. Α, οι πληρωμές δεν, αλλα... δεν αλλάξαν οι πληρωμές. Έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τις αναλήψεις υποχρεώσεων για να προετοιμαστούμε για την επόμενη χρονιά μόνο. Αυτό είναι. Οι πληρωμές δεν αλλάζουν. Ο Πρόεδρος, επιτρέψτε μου να εκφράσω την αμέριστη μου, τον αμέριστο θαυμασμό μου για τον κύριο Γκότμανες. Σα ευχαριστώ, λέει ο κύριος Γκότμανες. Όχι, εγώ σα εκφράζω τον θαυμασμό μου. Γιατί είναι πολλέ οι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ήλπιζαν και θα, είχαν, θα θεωρούσαν ιδιαίτερη τιμή το να έχουν ένα πρωθυπουργό ικανό και εργατικό και αποτελεσματικό όσο τον πρωθυπουργό, πρώην πρωθυπουργό κ. Γκοτμάνης της Λιθουανίας. Είναι τιμή για μας να έχουμε τέτοιου βεληνικούς μέλη. Outre, Πέρα του κυρίου Γκότμανης βέβαια, Α, όχι. Λε, Λετωνία, έκανα λάθος τη χώρα. <laughs> Με συγχωρείτε. Λάτβια, Λάτβια. Λάτβια, Λάτβια, λέει ο πρόεδρος. Λάτβια, Λάτβια, να μην μπερδευόμαστε. I am the bad boy. I am. No, no, Sorry, I'm so sorry. Ναι, εγώ βρίσκομαι έναν δίκο. Και λυπούμε. Λετωνία, Λάτβια. Ο εισηγητής λοιπόν. Προτείνει λοιπόν τις, με τις προφορικές του τροπολογίες και αν δεν ζητεί κανείς το λόγο, αυτό που προτείνω είναι να ψηφίσουμε το σύνολό του τον πίνακα αυτών με την προσαρμογή που αναφέραμε νωρίτερα, δηλαδή τη διαγραφή του, της γραμμής 19.01.04.04, δηλαδή της τροπολογίας 914 ή 227 για την ΚΕΠΑ. Και αν δεν έχετε αντίρρηση για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα λοιπόν, προτείνω συνολικά να ψηφίσουμε τον πίνακα ε, χωριστά μόνο τις χωριστές ψηφοφορίες που είναι ο μικρός πίνακας από κάτω στη σελίδα αυτήν. Συνολικά λοιπόν ο πίνακας, on block, ποιος είναι υπέρ του πίνακα και των προφορικών τροπολογιών. Κατά. Ένας. Ε, αποχές Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια κύριε ε, εισηγητά. Εγκρίθηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία η πρότασή σας. Και ευχαριστώ όλους που συμπράξατε σε αυτή τη διαδικασία που είναι και πολύ περίπλοκη αλλά και πολύ απλή ταυτόχρονα. Πάντως ασυνήθιστη. Με συγχωρείτε, πίνω και λίγο καφεδάκι για να αντέξω. Εάν ε, επιτρέπετε κύριε εισηγητά, εγώ προτείνω τώρα να κοιτάξουμε στις χωριστές ψηφοφορίες τι έχουμε. Πάλι στον ίδιο πίνακα, τη μονή αυτή σελίδα, όπου έχουμε στο κάτω σημείο ένα τετράγωνο, ένα παρελόγραμμο, με χωριστές ψηφοφορίες, οι οποίες αφορούν είτε τροπολογίες για το έγγραφο 10, όπως αναφέρεται άλλωστε, είτε για το έγγραφο 10 ΡΑΠ. Πρόκειται για τροπολογίες για τις οποίες ορισμένες ομάδες ζήτησαν ε, χωριστή ψηφοφορία προκειμένου να εκφράσουν θέση η οποία δεν είναι απαραίτητα ταυτόσιμη με αυτή του συγκητού. Έτσι ώστε να γίνει ψηφοφορία χωριστό. Τροπολογία 303 λοιπόν. Στο έγγραφο 10, 2 στη σελίδα 38. Γραμμή 18 020302 και ο κύριος Πόρτας, μέρους της Γκουε, η Γκουε μάλλον έχει στη συγχωριστή ψηφοφορία. Στο ελληνικό κείμενο είναι η σελίδα 36 επί των 82 του εγγράφου 10. 2. Κύριε Σιγητά, είστε υπέρ τροπολογίας. Ναι. Ο εισηγητής εμένει στην αρχική του θέση. Υπέρ δηλαδή. Υπέρ είναι ο εισηγητής. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Ο κύριος Πόρτας. Βεβαίως. Τρεις, και άλλοι δύο συνάδελφοι, δηλαδή τρεις κατά, αποχές δεν υπάρχουν. Εγκρίνεται ως εκ τούτου. Μετά έχω την τροπολογία, των προϋπο... την ε, τροπολογία προϋπολογισμών, Butch 9803, δεν ξέρω γιατί, έγγραφο 10 του εισηγητή. Το 10 RAP, Ένα μόνο τεύχος έχουμε εδώ. Στη σελίδα 38, γραμμή 180303. όπου η σοσιαλιστική ομάδα ζητάει χωριστή την ψηφοφορία για τα σχόλια. Για τα σχόλια, έτσι. Ο εισηγητής τι λέει. Ο εισηγητής θα είστε υπέστη της τροπολογίας και βέβαια αποδέχεται και τη χωριστή ψηφοφορία, δεν υπάρχει εμφολία. Καλώς. χωριστή ψηφοφορία ως προς τα σχόλια. Ποιος είναι υπέρ των σχολείων. Κατά μάιτρες παρακαλώ. Οι σοσιαλιστές προφανώς και κάποιοι άλλοι ίσως τάσσονται κατά των σχολείων. Ναι, πρέπει να ανάψουμε το κέντρο. Κίκο. 21 υπέρ. Κατά παρακαλώ. 14. Λοιπόν, λιγότερες λοιπόν είναι οι ψήφοι κατά. Εγκρίνεται η ψηφοφορία. εγκρίνεται η τροπολογία, εγκρίνονται μάλλον οι ε, παρατηρήσεις. Καλά μετρήσαμε ή ψήφισαν και Συμβούλιο και Κομισιόν μαζί με τους άλλους. Προχωρώ. Σελίδα, ε, τροπολογία 274. Επανέρχομαι δε στο έγγραφο 10, αλλά το τρίτο τεύχος αυτή τη φορά. Το κείμενο βρίσκεται στη σελίδα 3. 22, 01, 02, 11. όπου και πάλι η σοσιαλιστική ομάδα είναι εκείνη η οποία ζήτησε διαφορετικά σχόλια για το αποθεματικό. Ο εισηγητής πρόεδρε πρόκειται για ένα αποθεματικό για διαφορετικά πράγματα. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα. Ε, μπέρδεψα την ε, γραμμή. Μάλιστα, εδώ έχουμε αποθεματικό για το κοσποπέδιο. Ο εισηγητής θα είστε υπέρ του αρχικού κειμένου. Ποιο Ποιος είναι υπέρ τη τροπολογία μαζί με τι παρατηρήσει, μαζί με το αποθυματικό τη παρατηρήση. Εδώ θα είναι διαφορετική η έκβαση τη ψηφοφορίας. Αυτή τη φορά δεν θα ψηφίσει το Συμβούλιο, λέει ο πρόεδρο. 18. Qui est contre 18. Κατά παρακαλώ. Αχα. Αχαχα! Dix-neuf. 19 contre. Et donc l'amendement est rejeté. 19 κατά απορρίφεται η τροπολογία η αριστερά επεκράτησε της δεξιάς, κατήσχησε με κάποιες προδοσίες. Άρα το αποθεματικό καταργείται, έρεται, αποδεσμεύεται μάλλον. Ε, τώρα πάμε στο έγγραφο 10, τεύχος τρίτο, τροπολογία 290, στο κείμενο στη σελίδα 11. Πρόκειται για τη γραμμή 26010211. Με χωριστή ψηφοφορία στο αποθεματικό πρόκειται για τη σελίδα 12 στο ελληνικό κείμενο, επί των 48. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο. Α, γίνεται, γίνονται δύο ψηφοφορίες, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, και πάλι έχουμε αποθεματικό. Αυτή τη φορά το ΕΛΚ ζητεί χωριστή ψηφοφορία και έτσι ψηφίζουμε πρώτον το αποθεματικό της πρώτης παραγράφου. Αυτό είναι του Κωσόβου. Α, όχι, τέλειωσε το κοσμοπέδιο. Ούτε Λιθουανία είναι, ούτε Λετωνία είναι. Α, καταλήξαμε στις μελέτες εν τέλει. Σε τι μελέτες, τι μελέτες είναι αυτές. Α, δεν είναι γνωστό. Θα μας πει όμως η εισηγητής, θα μας πει ποια είναι η άποψή του. Ναι, είναι αυτό που ξεκίνησα νωρίτερα να εξηγώ. Αν θυμάμαι καλά, η σοσιαλιστική ομάδα είχε ζητήσει τη χωριστή ψηφοφορία, ήθελε μάλλον να ζητήσει τη χωριστή ψηφοφορία. Δεν υπάρχει αντίρρηση για τη γραμμή αυτή, δεν υπάρχει πρόβλημα έχουμε δύο ανεξάρτητα το ένα από το άλλο αποθεματικά. Το ένα αποθεματικό έτσι ώστε να προσδιοριστεί τι είδους μελέτες ε, αναπτύχθηκαν και πληρώθηκαν. Εδώ δεν έχουμε συμφωνήσει προς το αν είναι ε, ικανοποιητική η απάντηση Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Το δεύτερο, το αποθεματικό, έχει να κάνει με το αποθεματικό για την Όλαφ. Τη νομική τη βάση. Το πρώτο λοιπόν έχει να κάνει με το αν είναι ικανοποιητικέ οι μελέτες όπου θεωρεί ο συζήτης ότι χρειάζεται. Θα γίνει βέβαια η εξέταση και από την Επιτροπή και θα δούμε τα αποτελέσματα. Το δεύτερο, δεν θα ξαναστήσω όμως το λόγο και μετά, της Όλαφ, που θα θέλαμε να διατηρηθεί το αποθεματικό. Ο κύριος Κοτμάνης. στο έγγραφο 10, 26, 01, 11, για να δούμε πάλι τα νούμερα. Τελική, τελικό ποσό για τις πληρωμές είναι 5,6 εκατομμύρια ευρώ, 5 εκατομμύρια 600.000. Το ίδιο και στις αναλήψεις υποχρεώσεων. Σωστά κύριε Ισηγητά. Μάλιστα λέει ο κύριος Σόλια. Δεν επηρεάζεται το τελικό ποσό από τον τροπολογία Μόνο ένα κομμάτι από τα χρήματα αυτά πάει στο επαθηματικό. Πόσο μέρος όμως. Μερικά εκατομμύρια, δεν θυμάμαι. Ας το επαληθεύσουμε όμως. Στη σελίδα 12 θα το δείτε, λέει ο πρόεδρος. 3,7 και 1,8 εκατομμύρια. 1,867. Δεν χρειάζεται να το σας πω τα ψηλά. λέει ο κύριος Σίκτη. Ναι, σας το δώσω. That's all. That's all. Très bien. Très bien. Donc, y a deux... Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Ε, δύο διαφορετικά είναι τα αποθεματικά. Γιατί είχαμε ένα αποθεματικό μέχρι ότου λάβουμε περισσότερες πληροφορίες για τις δαπάνες που σχετίζονται με διάφορες εξωτερικές μελέτες, μελέτες που εκπονήθηκαν από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, για τις οποίες λάβαμε απαντήσεις ικανοποιητικέ. Σούριαν. Εξαρτάται από το πώς το κρίνει καθένα, ο καθένας. Εξαρτάται. Οι σοσιαλιστές θεωρούν ότι είναι ικανοποιημένοι, το ΕΛΚ θεωρεί ότι δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά του. Ο εισηγητής, προτείνει να διατηρηθεί το αποθεματικό. Μάλιστα. Και για το δεύτερο αποθεματικό που έχει να κάνει με την Όλαφ, όλοι συμφωνούμε να διατηρηθεί το αποθεματικό. Ωραία. Επομένως, στην πρώτη παράγραφο. Ο εισηγητής είναι υπέρ της διατήρησης του αποθεματικού και της τροπολογίας 290. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ της διατήρησης. 23. Κατά παρακαλώ. Πολύ λιγότερη. Διατηρείται λοιπόν το παθηματικό. Δεύτερη παράγραφος. Υπέρ της διατήρησης του παθηματικού νομίζω τάσεται η ευρύτερη πλειοψηφία της ομάδας της Επιτροπής κατά Α, όλοι θέλουν να διατηρηθεί. Αποχές, ομόφωνα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Άρα έχουμε διεκπαιρεώσει το πιο δύσκολο. Και τώρα έχουμε εγκρίνει τις προφορικές τροπολογίες. Έχουμε εγκρίνει τις τροπολογίες για τις οποίες έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία. Και τώρα προτείνω να ψηφίσουμε συνολικά, τον μπλοκ τις τροπολογίες δεύτερης ανάγνωσης, έκτος από αυτές που μόλις υιοθετήσαμε, που περιλαμβάνονται στο έγγραφο 10 ραπ. Ποιος είναι υπέρ των τροπολογιών αυτών. Σας ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. εγκρίνονται. Και εν τέλει, θα δούμε τον πίνακα υπαριθμών 10 που ανακεφαλαιώνει όλες τις τροπολογίες πρώτης ανάγνωσης που δεν τροποποίησαν οι πρόσφατες μας ψηφοφορίες, αυτές που κάναμε μόλις τώρα δηλαδή, αλλά που θέλουμε να επαναφέρουμε σε δεύτερη ανάγνωση. Ποιος τάσεται υπέρ αυτών των τροπολογιών στο σύνολό τους. Σας ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με την προηγούμενη ψηφοφορία. Λογικό και συνεπές ευχαριστώ τον, τον εισηγητή, τους συντονιστές και όλους τους συναδέλφους που ε, δέχτηκαν καταρχάς να ακολουθήσουμε αυτή τη ε, διαδικασία που ήταν τόσο απαραίτητη αλλά και κάπως δύσκολη ίσως ε, δημιούργησε κάποιες και προβλήματα προβλήματο ορισμένου. Δεν κλείσαμε όμω ακόμη τον προπολογισμό του 2010, γιατί τώρα έχουμε και την φιλολογία. Μετά τα νούμερα έρχεται η φιλολογία. Έχουμε δηλαδή το σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο παίρνουμε στα χέρια μας. Πάνω σε αυτό έχουμε μια σειρά τροπολογιών και κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες που θα μας ε, εξηγήσει ο εισηγητής όπως προχωράμε. Μήπως θα ήθελε ο εισηγητής να κάνει μία σύντομη παρουσίαση ή να δούμε τις τροπολογίες αμέσως. Κύριε Σούριαν, πρώτον νομίζω ότι οι ομάδες θα έχουν δουλέψει τα θέματα αυτά. Τα ξέρουν. Εγώ προσπάθησα στη γνωμοδότησή μου να ενσωματώσω τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις των συναδέλφων στο βαθμό του δυνατού. Δεν χρειάζεται πλέον, πιστεύω, να γίνει διεξοδική συζήτηση. Υπάρχουν κάποιες προφορικές τροπολογίες. Το κείμενο έχει διανεμηθεί και νομίζω μπορούμε να δούμε την κάθε τροπολογία με τη σειρά τη. Καλώς λέει ο πρόεδρο. Ας δούμε τώρα τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Έκθεση Φέρμ λοιπόν, μάλλον τροπολογία Φέρμ και Παλτζάνη ε, σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα, τι λέει ο συγητή. Ο συγητή είναι υπέρ. Α ψηφίσουμε λοιπόν το πρώτο κομμάτι. Κατά. Ουδή. Αποχέ. Ομόφωνα. Συγχαρητήρια στους συντάκτες. Δεύτερο τμήμα που ξεκινάει με το which might cause που θα μπορούσε να προκαλέσει ο εισηγητής. Είναι κατά υπέρ παρακαλώ. Καταμέτρηση. Ε, ο κύριος αν δεν 20 χέρι ξυνότανε, αλλά να το μετρήσουμε. Εντάξει, 16. Κατά. Κατά. Λουκ είπα, κατά. Α, κατά είσαι. Δεκαεπτά. Α, όχι, 16 υπέρ, 17 κατά. Μάλιστα, απορρίπτεται λοιπόν η τροπολογία με την ψήφο του Ζαλεκ Πάμε στην παράγραφο 3. Έχουμε προφορική τροπολογία εδώ. Α, θέλω να μας το παρουσιάσει όμως αυτό ο κύριος εισηγητής μας. Δυστυχώς χωρίς μικρόφωνο. Ε, Μάλιστα. Θα ήθελα να προτείνω μια μικρή αλλαγή Υπάρχουν εδώ διάφοροι υπολογισμοί. Σε πόσες φορές αλλάξαμε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχω δει και τρία και τέσσερα και πέντε να γράφει. Και θα πρότεινα για να απεφύγουμε οποιαδήποτε συζήτηση και να στείλουμε ακόμα πιο ηχηρό μήνυμα να πούμε. Θυμίζει ότι από το 2007 η Δημοσιονομική Αρχή επανειλημμένα υποχρεώθηκε να αναθεωρήσει. Εντάξει, για να μην πούμε ακριβή αριθμό 3, 4 ή 5, να πούμε ότι υποχρεωθήκαμε εμείς να αλλάξουμε επανειλημμένα. Αυτό λέει ο κατάλογος ψηφοφορίας που μας έχει δυναμηθεί. Ναι. Μπορούμε να ε, αφαιρέσουμε στο τέλος, όπως βλέπετε επίσης που λέει, ε, απρόβλεπτες or unforeseen. Με αυτές τις αλλαγές ψηφίζω. Θέλετε να αποσύρετε το or foreseen. Όχι, or unforeseen, ε, τις απρόβλεπτες. Αυτό θέλετε να το αποσύρετε. Να πούμε επανειλημμένος και όχι δύο, τρεις ή τέσσερις φέγορες. Α, όχι, διορθώνει κύριε Σούριαν. I misunderstand the typing. Α, δεν έβγαζα τα γράμματα. Ναι. Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια. το ακριβές κείμενο είναι αυτό που αναγράφεται στον κατάλογο ψηφοφορίας. Ζητώ συγγνώμη. Εγώ είχα ένα άλλο έγγραφο του Ουγγρικού Κοινοβουλίου υπόψη μου και ε, ε, είχα μπερδευτεί. Ωραία, καλώς λέει ο Πρόεδρος. Πάντως, Μπορεί να μείνουν ίσχυοι βουλευτές γιατί η προφορική τροπολογία ανταποκρίνεται απόλυτο σε αυτό που γράφει ο κατάλογος ψηφοφορία. Μου προκαλεί ευθυμία γιατί μέχρι τελευταίο ευρώ μπορούμε να ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε για κάθε μελέτη, αλλά δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε από το 2007 μέχρι σήμερα πόσες φορές αλλάξαμε τη διοργανική συμφωνία. Είναι αρκετά ε, αστείο αυτό. Λοιπόν, υπέρ, ευχαριστώ. Κατά, κανείς, αποχές, εγκρίνεται. Καλώς. Η τροπολογία υπαριθμών 4 τώρα. Υποθέτω ότι θέλει και εδώ ο εισηγητής να μας παρουσιάσει την προφορική τροπολογία. Οριζόντια λέει εδώ και προφορική. Ναι, ναι, Πρόεδρε. Εχθές στη συνεδρίαση των συντονιστών συμφωνήσαμε για μια τροπολογία που να λέγει ότι τροποποιείται η ε, τροπολογία 4 με τον τρόπο που αναγράφεται εδώ στον κατάλογο με προσαρμογή, αναθεώρηση και επαλήθευση της ε, περίοδου 2007-2013 συμπεριλαμβανομένης της παράτασης μέχρι το 2015-2016. Πρόκειται για μία έκθεση, μια επανάληψη μάλλον της παλιάς διατύπωσης που είχε και έκθεση κυρία Γικιά. Ότι έχουμε τρία βήματα. Ένα προσαρμογή, ε, επαλήθευση και αναθεώρηση. Και στη συνέχεια θα ζητήσω και άλλη αλλαγή αν εγκριθεί αυτή. Δηλαδή, θέλετε να ψηφίσουμε πρώτα την οριζόντια τροπολογία, μετά την προφορική. Τώρα θα σας πω για την οριζόντια. Το κείμενο που κατέθεσαν οι σοσιαλιστές συνάδελφοί μας έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει το Α και το Β ε, μόλις αναλάβει. <laughs> Και στη συμφωνία που ζητούμε ε, να χρησιμοποιήσουμε άλλη διατύπωση, όχι μόλις αναλάβει, το συντομότερο δυνατόν. Μόλις αναλάβει με το καλημέρι σας την άλλη μέρα αυτό θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Αλλά εντάξει να τη πιέσουμε χρονικά να πούμε το συντομότερο. Νομίζω ότι είναι καλή αυτή η συμφωνία. Και αυτό το κείμενο όπως βλέπετε είναι στην τροπολογία 4, 12, 17, 25 και 32. Ε, ψηφίζοντας άπαξ θα κάνουμε αυτές τις αλλαγές σε ε, όλες τις τροπολογίες ανεξάρτητα από το αν αυτές πλέον εγκριθούν ή όχι. Μάλιστα λέει ο Πρόεδρος. Οπότε Κάνουμε μία διάκριση εδώ στην τροπολογία υπαριθμών 4. Έχουμε δύο διαφορετικά προβλήματα και δύο διαφορετικές υποδείξεις του εισηγητού. Θα ψηφίσουμε πρώτα την πρώτη αλλαγή και μόνο, την προφορική του τροπολογία που συνίσταται ε, και αφορά την τροπολογία 4 και σε περίπτωση που εγκριθούν τη 12, 17, 25 και 32 να μην πούμε από την πρώτη μέρα μόλις αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθήκοντα, αλλά το συνομοτέρο. Δύο ζητούν το λόγο γι' αυτό, ο Γιώραν. Συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα από αυτού. Ως παλιός δημοσιογράφος όμως είμαι λίγο ευαίσθητος πάντα με τη διατύπωση. Θα πρέπει να λέμε μία προσαρμογή, μία αναθεώρηση και μία επανεξέταση δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ίδιο άρθρο, είναι θέμα άρθρων στην αγγλική. Ε, εν και τι θα χρησιμοποιούμε. Αυτή είναι η δεύτερη προφορική τροπολογία, την ε, σημειώνουμε και υπάρχουν ε, και <coughs> αγγλομαθείς ε, γλωσσολόγοι, αγγλόφωνοι, οι οποίοι θα είναι ικανοποιημένοι. Συγγνώμη, δεν μπόρεσα να είμαι παρούσα εχθές στη συνεδρία των συντονιστών, Αλλά έχω μία παρατήρηση επί της ουσίας. Επανειλημμένως το έχουμε ψηφίσει αυτό στο Κοινοβούλιο, καθώς επίσης ε, και μία παράταση του 50 και του 60, αλλά θα ήθελα να γίνει κατά τμήματα ψηφοφορία για να μπορέσω να το καταψηφίσω. Όπως το ανταλαμβάνομαι εγώ, θα μπορούσε να είναι μεν μία επιλογή, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι για το 2015, 2015 και 2016 και δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, συμφωνούμε. Έτσι κι αλλιώς δύο χωριστές ψηφοφορίες θα κάνουμε, είναι διαφορετικά τα προβλήματα. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε πρώτα την οριζόντια λεγόμενη τροπολογία για να πούμε το συντομότερο δυνατόν. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Με δύο ψήφους κατά. Αποχές και χωρίς αποχές εγκρίνεται. Καλώς. Έχω την αίσθηση ότι κάποιος παρόν στην αίθουσα έχει μάλλον ανακουφιστεί από την ιδέα αυτή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δράσει το συντομότερο και όχι από την ανάληψη των καθηκόντων της ίδια μέρα. Έτσι. το λέω απλώ Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη τροπολογία, την προφορική, ε, για αυτό που πρότεινε ο Ράιμερ Μπέγκερ και που οι φιλελεύθεροι ζήτησαν χωριστή ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ αυτής της προφορικής τροπολογίας. Κυρία Γένσεν, μπορούμε να έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο, το πρώτο. Α, το, ε, χωριστή τη χωριστή θέλετε. Ωραία. Ναι, ναι, αυτό θέλουμε. Ε, το πρώτο τμήμα με την προσαρμογή, αναθεώρηση και επανεξέταση κτλ. Ε, του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και μετά το επόμενο τμήμα συμπεριλαμβανομένης παρατάσεως μέχρι το 2015-2016. Μάλιστα. Η χωριστή της χωριστής ψηφοφορίας, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα μέχρι την περίοδο 2007-2013, μέχρι εκεί Τελεία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Χωρίς αποχές εγκρίνεται με δύο ψήφου κατά. Λοιπόν, το δεύτερο τμήμα τώρα, συμπαραμβανωμένες παρατάσεις μέχρι το 2015-2016. Υπέρ. Κατά. Δύο ομάδες είναι κατά. Άλλα είναι μικρές και δεν μπορούν να εμποδίσουν την έγκριση... Α, τρεις ομάδες, συγγνώμη. Όχι, αποχή η τρίτη ομάδα. Α, αποχή, συγγνώμη. Γκουε, αποχή. Λοιπόν, αυτό το τμήμα της προφορικής τροπολογίας εγκρίνεται επίση. Σας ευχαριστώ. Ε, είναι λίγο μακροσκελής η διαδικασία. Είναι περίπλοκο και θα πρέπει να προχωρούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, Ερχόμαστε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 5 των σοσιαλιστών. Και εδώ έχουμε προφορική τροπολογία. Και ψηφοφορία κατά τμήματα. Κύριε Σιγητά μου. Ε, Κύριε Πρόεδρε, αποσύρω την πρόταση για την κατατμήματα ψηφοφορία. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μία προφορική τροπολογία στο κείμενο που λέει ότι η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση θα αντικαθίσταται από τη διαδικασία των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών και αυτά θα γίνει στα πλαίσια του επόμενου πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου και με την προφορική αυτή τροπολογία θα ήθελα να υποστηρίξω το σύνολο της τροπολογίας. Σας ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται λοιπόν κατά τμήματα εδώ ψηφοφορία ο εισηγητή για την προφορική τροπολογία και κανεί άλλο δεν το ζητεί. Ωραία. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία όπω τροποποιήθηκε. Κατά. δύο αποχέ ομόφωνα. Αρκετά σπάνιο για αξιοσημείο του. Ερχόμαστε τώρα στις τροπολογίες της κυρίας Κτρούπελ. Ο εισηγητής ε, κατά το Αυτό δεν είναι συνάδει με όλα όσα έχουμε ψηφίσει μέχρι τώρα. Επομένω, νομίζω ότι θα πρέπει να καταπέσει αυτή η τροπολογία. Κύριε Σιγητά, εσεί τι νομίζετε, καταπίπτει. Ναι, όντω. Η τροπολογία καταπίπτει. Διότι δεν συνάδει με όσα έχουμε πει, δεν θα την υποβάλουμε σε ψήφισμα. Καταπίπτει. Επτά. Τι λέει ο μα. Είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πούμε στη Χέλγα ότι η απουσία της μια ενθουσιώδης ομοφωνία επικράτησε για την επτά. Ε, τροπολογία 8 ψήφι υπέρ. Κατά. Α, δεν έχουμε κατά. Πέντε. Αποχές, χωρίς αποχές, Εγκρίνεται όμω η πλειοψηφία ήταν υπέρ. Στην παράγραφο 11 έχουμε δύο τροπολογίε. Πρώτα μία του κύριου Πόρτα. Ο εισηγητής είναι αντίθετος, ψήφι υπέρ. Υπέρ ο κύριος Πόρτα. Κατά. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι αντίθετη, απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 10 του Γιώργαν Φέρμ και της κυρίας Μπαλτσάνη. Η προφορική τροπολογία του εισηγητού μας. Παρακαλώ. Ναι, προτείνω να σκεφτούμε όχι μόνο το σημείο 3 αλλά και το σημείο 23 όπως είναι στην ε, τροπολογία αλλά θα ήθελα να συμπεριλάβουμε και τα σημεία 21 και 22. Πρόκειται για μια προφορική τροπολογία η οποία συνάδει με όσα έχουμε ψηφίσει στην παράγραφο 3α νέα, διότι μιλάμε Adjustment Review Revision, επομένως ε, αυτά αντιστοιχούν στα διάφορα άρθρα 21, 22 και 23. Ποιος είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας, ως τροποποιήθηκε με την προφορική τροπολογία του εισηγητή. Κατά, κανείς, αποχές, απέχεται, δύο αποχές. Εγκρίνεται, σας ευχαριστώ. Τροπολογία 11. Από τον κύριο Λαμασούρ. Η τροπολογία για την νομική συνέχεια που σας παρουσίασε εχθές. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας του Προέδρου. Je Σας ευχαριστώ. Κατά. Κυρία Σεν, είστε αφηρηκτοί. επιμένει να εκφράζει την άποψή της. Κατά, κανένας. Ευχαριστώ τους πάντες εκτός μίας. Εγκρίνεται λοιπόν 12 των σοσιαλιστών. Εδώ ισχύει η οριζόντια τροπολογία, αλλά ποιος είναι υπέρ της 12. Ο εισηγητής είναι κατά. Πρέπει να μετρήσουμε. 8, 9, 10, 11, Non, 11, 12, 13. Donc c'est la gauche dure. αριστερά euh, Madame Συν την ομάδα της κυρίας Ανδρέασεν. Πόσους έχουμε δηλαδή? Vous Monsieur 14. 14. Ο Ζανλούκ Μποντεάν δεν κουνήθηκε. Κατά. Λοιπόν, απορρίπτεται. Τροπολογία, παράγραφος 13. Η Έλγα για την τροπολογία 13. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Δύο αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14, η οποία συμβατεί με τη 13 της κυρίας Γένσεν. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Μπόλικη. Κατά. Μία. Αποχές. Καμία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14. Τροπολογία. Γκρέσλε. Συμφωνεί και ο εισηγητής. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Δύο κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15. Καταρχάς, μία ε, τροπολογία της κυρίας Γένσεν. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ένας κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17, που είναι συμβατή με την τροπολογία 16 και που φυσικά θα επωφεληθεί και από την οριζόντια τροπολογία. Ο εισηγητής δεν ε, είναι σύμφωνος. Ποιος είναι υπέρ. Η σκληρή αριστερά και πάλι. Says. 16. Κατά. 18. 18 κατά, που είναι λοιπόν παραπάνω των 16 που ήταν υπέρ, απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Γκρέσλε. Υπέρ. Ευχαριστώ. Ποιος τολμά να είναι κατά. Η κυρία Ανδρέασαν και η φιλελεύθερη είναι κατά. Αποχές. Μία αποχή. Και επομένως εγκρίνεται. 19 της Χέλγα Τρούπελ συμβατεί με την 18. Η είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ένας κατά. Αποχές και μία αποχή εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην παράγραφο 18. Τροπολογία 20 της Χέλγα Τρούπελ. η οποία τροποποιείται με μια προφορική τροπολογία του εισηγητή μας, ο οποίος θα ήθελε να εκφράσει την έκπληξή του. Κύριε Σιγητά, κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι μπορείτε να τη διαβάσετε, είναι γραμμένη και θα ήθελα με την αλλαγή αυτή να την υποστηρίξω. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας, της Χέλγια Τρούπελ, ως τροποποιήθηκε από την προφορική τροπολογία του συγητή, υπέρ. Αυτή η εικόνα είναι φωτογραφία των συντονιστών του ΕΛΚ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18α νέα. Τροπολογία 21 του κυρίου Χάγκλουν. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 της Χέλγια Τρούπελ. Ο εισηγητές είναι κατά. Υπέρ. Η σκληρή αριστερά και πάλι κατά. Η πλειοψηφία είναι κατά. Είναι σαφές, επομένως απορρίπτεται. Παράγραφος 21, δύο τροπολογίες, 23 του κυρίου Πόρτας. Ο εισηγητής είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. Για την τροπολογία του κυρίου Πόρτας. Ο κύριος Πόρτας είναι υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία είναι κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. Απορρίπτεται. Η 24 της Έλγα Τρούπελ, η οποία πρέπει να ψηφιστεί γιατί δεν ψηφίστηκε 23, αλλά ο εισηγητής είναι και πάλι κατά. Υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία είναι κατά. Απορρίπτεται. Παράγραφος 22, τροπολογία 25 των σοσιαλιστών, η οποία άπτεται και της οριζόντιας τροπολογία. Ο εισηγητής δεν τη θέλει. Υπέρ. Έχουμε λίγο παραπάνω από τη σκληρή αριστερά. Ça doit faire 13. 14. 14 pour. 14 υπέρ. Ποιο είναι κατά. Probablement un petit peu plus. 21. 21 κατά, Επομένω απορρίπτεται. Παράγραφο 24, έχουμε και πάλι τροπολογία του κυρίου Πόρτα. 26, υπέρ. Ο εισήγητή είναι κατά. Υπέρ, το fan club του κύριου Πόρτας. Σας ευχαριστώ. Κατά. Η πλειοψηφία είναι κατά. Λυπάμαι αγαπητοί συνάδελφοι. Περνάμε τώρα στην 27. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ της 27. Ευχαριστώ. Κατά. Δύο κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Εγκρίνεται. Παράγραφος 26. Τροπολογία 28. Υπέρ. Ο εισηγητή είναι κατά. Η φιλελεύθερη είναι και αυτή υπέρ, επομένως πρέπει να μετρήσουμε. 19 υπέρ, κατά. Combien 15. Donc cette fois 15. Εγκρίνεται λοιπόν αυτή η τροπολογία. Να συγχαρούμε τους συντάκτες. Παράγραφος 26. Δεν υπάρχει τροπολογία, αλλά ο εισηγητής ζητά κατά τμήματα ψηφοφορία. Για το πρώτο τμήμα ο εισηγητής είναι υπέρ. Όχι για να ακούσουμε τον συζητή. Micro, micro, Mr. I think... Νομίζω ότι είναι ψευδής αυτή η κατατμήματα ψηφοφορία. Η Επιτροπή δέχτηκε να μην ε, συμπεριληφθεί η παράγραφος 26. Αυτή ήταν ε, η πρότασή μου, να κρατήσουμε μόνο το δεύτερο τμήμα, γι' αυτό και είχα ζητήσει κατά τμήματα ψηφοφορία, αλλά η Επιτροπή αποφάσισε διαφορετικά. Άρα η παράγραφος 26 διαγράφεται. Επομένως, η τροπολογία καταπίπτει, αλλά η παράγραφος μένει. Όχι, ανάποδα. Η παράγραφος εξαφανίστηκε, άρα δεν υπάρχει λόγος για τροπολογία. Δεν μπορούμε να κόψουμε στα δύο κάτι που δεν υπάρχει. Bien. Bien. Là, on suit. Ωραία. Το πιασα τώρα. Παράγραφος 28. Τροπολογία 29. Ο εισηγητής είναι κατά. Και η φιλελεύθερη. Ποιος είναι υπέρ. Και πάλι σκληρή αριστερά. Κατά. Οι υπόλοιποι. Αποχές. Επομένως απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Και ο εισηγητής είναι κατά. Αλλά αυτή τη φορά η φιλελεύθερη είναι υπέρ. Επομένως πρέπει να μετρήσουμε. Ποιος είναι υπέρ. Δεκαεπτά υπέρ. Ποιος είναι κατά. jean κατά είμαστε εμείς. 18. με τον Jean-Luc. Και με την κυρία Αντρέασεν. Η οποία διαδραματίζει ρόλο κλειδί. Και δεν μ' αρέσει πάντα, αλλά τι να κάνω. Τέλος πάντων, ας μην το κάνουμε προσωπική υπόθεση τώρα αυτό, απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 31. Ingeborg Γκρέσλε, ο εισηγητής είναι προφανώς υπέρ. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Δύο κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Εμπλουτισμένη από την προφορική τροπολογία. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Πρέπει να το επισημάνω αυτό. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ένας, δύο κατά αποχές, καμία αποχή, εγκρίνεται. Παράγραφος 30. Δύο τροπολογίες εδώ. Η μία αποκλεί την άλλη. Τροπολογία 33. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Η αριστερά μόνο. Κατά. Οι υπόλοιποι αποχές, επομένως απορρίπτεται. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε τη 34. Ο εισηγητής είναι υπέρ της 34, αλλά Βλέπω ότι υπάρχουν και κάποιοι που είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ λοιπόν τη 34 της κυρία Τρούπελ. Η σκληρή δεξιά υποστηρίζει τη Χέλγα. Ça fait combien Non, mais il faut compter Γραμματεία κοιμάται μου φαίνεται, δεν μετράει καλά. Σεζ, και κόντρ. Δεκαέξι, κατά. 18. 18 κατά. Επομένως, απορρίπτεται. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια έχουμε δεν καταπίπτει 35 γιατί δεν πέρασε η 33, επομένω ψηφίζουμε την 35 του κυρίου Πόρτα. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Η αριστερά. Κατά οι υπόλοιποι. Επομένως, απορρίπτεται. Παράγραφος 31. Δύο τροπολογίες ασύμβατες μεταξύ τους. Η 36. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Λίγο παραπάνω από την αριστερά είναι και η κυρία Ανδρέας εδώ και ο κύριος Μοργκάντη που την υπερψηφίζουν. 13 pour. υπέρ, ποιος είναι κατά. Η πλειοψηφία είναι κατά. Ευχαριστώ. Επομένως απορρίπτεται και επομένως μπορούμε να ψηφίσουμε την 37. Ο εισηγητής την πιστεύει. Είναι υπέρ της τροπολογίας της κυρίας Γένσεν. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Μία αποχή εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπότιτλος πριν από την παράγραφο 33 ε, ο κύριος Μάνκα είναι αντίθετος, ο εισηγητής είναι υπέρ, ποιος είναι υπέρ, κατά, ευχαριστώ, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 38 της κυρίας Τρούπελ. Ο εισηγητής θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. να την υποστηρίξω την ε, τροπολογία 38 της Χέλκε Τρούπελ και υπήρξε και αίτημα από την ομάδα των συντηρητικών εχθές να κατατεθεί μια τροπολογία ως προσθήκη στην παράγραφο αυτή. Και τους υποσχέθηκα για να τηρήσουμε την παράδοση οι προφορικές τροπολογίες σε αυτή τη φάση να κατατίθεται από τον εισηγητή. Αυτό είναι άγραφος νόμος, δεν είναι επί χάρτου, αλλά είναι η παράδοση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και δεν θα ήθελα φυσικά εδώ να παραμελήσω την προφορική τροπολογία μιας ομάδος, θα την καταθέσω. Όσον αφορά στο περιεχόμενο όμως, έχω πολλές επιφυλάξεις. Νομίζω ότι δεν ε, συνάδει με το πνεύμα της συμφωνίας κυρίων να ζητάμε από όλους, από όλα τα θεσμικά όργανα να έρχονται εδώ και να μας εξηγούν τι δουλειά πρέπει να κάνουν, ποια είναι τα καθήκοντά τους. Γι' αυτό και με όλο το σεβασμό προς τους συντηρητικούς, το ε, περιεχόμενο δεν μπορώ να το στηρίξω ηγητής. Θα ήθελα όμως να ψηφιστεί και να δοθεί το δικαίωμα σε όλους να αποφασίσουν επί του θέματος αυτού. Ουσιαστικά σας ζητώ κατά τμήματα ψηφοφορία ή να ψηφίσουμε πρώτα την προφορική τροπολογία, αν τη δεχτούμε να την απορρίψουμε και κατόπιν ε, η υπόλοιπη τροπολογία υποστηρίζεται από τον εισηγητή. Πολύ ωραία, ευχαριστώ τον εισηγητή, διότι παίζει δίκαια το παιχνίδι. Η τροπολογία σας έχει διανεμηθεί, την έχετε, αλλά να δώσω φυσικά το λόγο στον ε, James Έλλης. Ευχαριστώ. Εχθές υπήρχε το πνεύμα ότι δεν είναι ο εισηγητής ε, να ζητήσει από τους γενικούς γραμματείς να έρθουν να εξηγήσουν. Εμείς θέλουμε όμως ε, να έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχει οικονομία στη διαχείριση των πολιτικών τους. Διότι αυτό σχετίζεται με μία άλλη τροπολογία του κυρίου Μάνκα, είναι η τροπολογία 40, στην οποία αναφερόμαστε στην ανάγκη να έχουμε νέα, και αυτό είναι ε, στο παράρτημα 4 για τα νέα στοιχεία, αλλά εκεί έχουμε και την οικονομία, αλλά η οικονομία δεν αναφέρεται εδώ. Η τροπολογία λοιπόν η προφορική τροπολογία είναι μια επενθύμηση στην Επιτροπή Προπολογισμών να έχουμε και το θέμα της οικονομίας ε, και όπως έχουμε και την αντίστοιχη δυνατότητα και στα νέα τιμάτα Ωραία. Έχουμε το κείμενο της προφορικής τροπολογίας χωρίς την εξήγηση, μας την παρουσίασε και ο εισηγητής, μας εξέφρασε και τις επιφυλάξεις του επί του περιεχομένου. Να ψηφίσουμε πρώτον την ε, προφορική τροπολογία που συμπληρώνει την τροπολογία 38 και κατόπιν να ψηφίσουμε την τροπολογία 38. Ποιος είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας που κατέθεσε ο εισηγητής. Ο εισηγητής είναι κατά. Ψήφι υπέρ. προφανώς. Ο κύριος Μπέγκε και η Σιδονία. Πολύ είναι υπέρ. C'est un amendement cross είναι γκάσια διακομματική τροπολογία. Ευχαριστώ. Και η Γκουε. Η Γκουε έρχεται να συνδράμει τους Βρετανούς συντηρητικού. Μα καλά, ζούμε εδώ στιγμές ε, εφορίας ε, θαυμάσια. Κατά. Η κατά είναι περισσότερη. Κρίμα. Δεν πειράζει. Καλό ήταν να γίνει αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, έτσι, αυτή η προσθήκη απορρίπτεται, αλλά θα θέσω σε ψηφοφορία την αρχική τροπολογία 38 της κυρίας Τρούπελ. Ο εισηγητής είναι υπέρ, άλλη υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Ο Τζέμις Σέλς υπερψήφισε την τροπολογία της κυρίας Τρούπελ, πολύ σπορτίφ, παρόλο που δεν είχε γίνει δεκτή η δική του προσθήκη. Και ερχόμαστε στην τροπολογία υπαριθμών 39 των σοσιαλιστών η είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ομόφωνα. Η τροπολογία 40 του κύριου Μάνκα. Εισηγητής είναι υπέρ. Ψήφι Κατά. Με δύο ψήφους ε, κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 41 του κύριου Πόρτας. Ο Συγητής δεν είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. το fan club του, οι οπαδοί του που υπεβαίνουν την γοέλα δεν είναι αρκετοί. Ναι, όντω. Απορρίπτεται. 42 ε, του κύριο μάνκα, είπε. Κατά. Αποχέ. Με δύο Μην Εγκρίνεται. Και τέλο η τροπολογία υπαριθμό 43 του κύριου μάνκα. Εξ ονόματο των σοσιαλιστών πλέον δεν είναι προσωπική του τροπολογία. Ψήφι κατά αποχές χωρίς αποχές εγκρίνεται ομόφωνα. Και τέλος, το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε, ψήφι υπέρ παρακαλώ, σας ευχαριστώ, κατά, με δύο ψήφους κατά αποχές και μία αποχή της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ πολύ όλα τα μέλη και όλος ιδιαιτέρως φέρνουμε ε, τους συνεργάτες μας. Δεν τελειώσαμε όμως με τη δεύτερη ανάγνωση εδώ. Έπεται η Ολομέλεια. Τώρα θα κληθούμε να πείσουμε τις πολιτικές μας ομάδες να ακολουθήσουν ε, και να υπακούσουν στη σοφία της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ κύριε Σίγητα για τις προτάσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε και άλλη ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό. Το σημείο 9 για την έκθεση του Ράιμερ Μπέργκε. και πρόκειται για τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας. Είναι η λογική συνέχεια και είμαι υποχρεωμένος να κάνω χωριστή ψηφοφορία γι' αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα είναι και η ίδια ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ για να είμαστε και συνεπείς τα όσα ψηφίζουμε. Όλοι, οι πάντες, όλοι ψηφίσατε σε βασιλετός κατά, οι ίδιοι αποχές, οι ίδιοι. Ακριβώ ταυτόσιμη λοιπόν η ψηφοφορία και σα ευχαριστώ. Το ίδιο ισχύει και για το 10, κινητοποίηση του μέσου ευελιξία. ο Ράιμερ Μπέργκερ Μα προτείνει ε, αυτό, ο εισηγητή είναι υπέρ, οι ίδιοι υπέρ, οι ίδιοι κατά, υποθέτω, είναι συνεπεί με τον εαυτό του, αποχέ τα ίδια το αυτόν Για το 11. Α, εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουμε εντελώ θέμα. Θα περάσουμε στο διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 10 του 2009 αλλά συνδέεται και με το προηγούμενο. Δεν Καλά είπα ότι αλλάζουμε θέμα, δεν εννοώ αυτό ακριβώς. Ε, παραμένουμε βεβαίως στο προϋπολογισμό και στο πακέτο για τη χρηματοδότηση του 2010 παίρνουμε πιστώσεις ε, πληρωμών ε, από το 2009 για να χρηματοδοτήσουμε το σχέδιο ανάκαψης. Αποουσιάζει η Γιούτα Χάουκ, θα μας τα πει ο Γιώραν Φέρμ, είναι ήδη... Όχι, θέλει το λόγο. Θέλει το λόγο πριν ψηφίσουμε. Παρακαλώ, κύριε ε, αναπληρωτή εισηγητά. Ναι, η Γιούτα Χάουκ ζητά συγγνώμη, είναι στην Αφρική αλλά μου ζήτησε να σας παρουσιάσω μία επεξηγηματική της δήλωση, διότι υπάρχουν ε, κάποια πράγματα τα οποία είναι τελείως τεχνικά και κάποια άλλα, όπως είπατε κι εσείς, συνδέονται άμεσα με τη συμφωνία που είχαμε στη συνδιαλλαγή, διότι είναι τμήμα του προγράμματος ανάκαμψης, αλλά θέλει να επισημαίνουμε και κάποια σημεία τα οποία θεωρεί ότι είναι ε, προβληματικά και θα πρέπει να τα δούμε. Παραδείγματο χάρη, ζητούν, μα ζητούν να επιστρέψουμε 3,4 δι ευρώ στα κράτη-μέλη διότι δεν έγιναν πληρωμές σε κάποιες τομείς. Και η εισηγήτρια θέλει να κατανοήσουμε ότι επικρίνει απόλυτα τις ε, έλλειψες πληρωμής για τα 1, 2 ε, και 4 και επίσης η αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων ήταν κάτι το οποίο ήθελε το Κοινοβούλιο στο προϋπολογισμό πέρσι αλλά δεν το υλοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει λοιπόν να το εξετάσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει την απόδοσή της στην εφαρμογή των αποφάσεων των δημοσιονομικών αρχών. Και αυτό είναι το βασικό και νομίζουμε ότι είναι ένα από τα θέματα στα οποία θα πρέπει να επανέλθουμε πάρα πολύ σοβαρά εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμών και όχι μόνο στη διαδικασία του προπολογισμού. Θα πρέπει να αρχίσουμε να το συζητούμε εκ των προτέρων για του χρόνου. Και αυτό είναι ένα από τα μηνύματα της συγγήτριας. Επίσης, επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσουμε με τη διαδικασία πλούστευσης, ώστε να πλουστευθούν οι δαπάνες. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα τα οποία θα ήθελα να τονίσει. Ωστόσο, δεν έχει άλλη επιλογή παρά να μας ζητήσει να δεχθούμε αυτό το σχέδιο κειμένου και επομένως προτείνω να το υπερψηφίσουμε παρά τις επικρίσεις της. Ευχαριστώ Γιώργο για αυτή τη σημαντική διευκρίνηση και όσα μας είπατε ονόματος της Ιούτα Χάουκ. Με πολύ μεγάλη προσοχή σας άκουσαν οι ε, σημερινοί και επόμενοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ παρόντες. Ο Τζέιμς ζήτησε το λόγο από αυτό. Θα θέλω να αφαιρθώ σε κάτι που είπε Γκέρεν για την εφαρμογή του προπολογισμού. Προφανώς εδώ έχουμε τα 3,4 δισεκατομμύρια που δεν έχουν ε, εκτελεστεί, αλλά από την Επιτροπή και την εμπειρία μου που έχω σχέση με αυτού, βλέπω ότι πολλές φορές υπάρχουν κανόνε δημοσιονομικοί οι οποίοι παρεμβαίνουν στον ε, δημοσιονομικό όγκο ε, κατά τρόπο μαζικό και νομίζω ότι μια και εδώ η κυρία Γκρέσλε μπορούμε να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιούνται οι, νέοι αυτοί, οι κανονισμοί αυτοί ε, από εδώ και μπρος. γιατί πρέπει εφόσον υπάρχει βέβαια ο δημοσιονομικός έλεγχος, εκείνοι οι οποίοι έχουν τη διαχείριση των ε, κονδύλιων αυτών να μπορούν να εφαρμόζουν, να εκτελούν τα ποσά αυτά ελεύθερα. Βεβαίως, λέει ο πρόεδρος, έχετε απόλυτο δίκαιο. Πρόεδρε, πολύ σύντομα ως εισηγητής για τον προϋπολογισμό θα ήθελα να σημειώσω ότι ε, υποστηρίζουμε την πρόταση για υλοποίηση στο στάδιο αυτό. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι για το θέμα που ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές, νομίζω ότι χρειάζεται λεπτομερής ανάλυση. Υπάρχουν κάποιες φιλοδοξίες μερικές φορές από πλευρά των βουλευτών να δίνουν όντως περισσότερα κονδύλια, χωρίς όμως να γνωρίζουμε το ευρύτερο πλαίσιο. Ίσως είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι. Υπάρχουν ορισμένε άλλε περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν είναι τόσο φιλόδοξη ω προς την εκτέλεση. Και εκεί μπορούμε πράγματι να πούμε ότι η Επιτροπή πρέπει να διαχειρίζεται αυτό το οποίο, στο οποίο έχει συμφωνήσει η Δημοσιονομική Αρχή. Αυτό το δεύτερο σενάριο. Και το τρίτο που ανέφερε και ο James είναι ότι υπάρχει καλή πρόθεση από την Επιτροπή και η φιλοδοξία από τη Δημοσιονομική Αρχή, αλλά σε τεχνικό επίπεδο οι λεπτομέρειες μας δυσκολεύουν πολύ τη ζωή. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε πέρα. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Ρεαλισμό στις φιλοδοξίες μας, να πιέσουμε την Επιτροπή για την εφαρμογή και να αλλάξουμε τους κανονισμούς όπου αυτό χρειάζεται. Είναι καλό νομίζω το καλό αυτό για την επόμενη χρονιά. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, ξέρετε τι παρατήρησε από πλευρά του Σκιώδους, ξέρετε ότι ο Λάσλο ήρθε μαζί με τη σκιά του σήμερα. Με αυτές λοιπόν τις παρατηρήσεις, που είναι πολύ σημαντικές, υπέρ. Κατά. Είστε κατά. Κατά είσαστε. Μάλιστα, καλώς. Αποχές. Χωρίς αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Και τώρα, αν δεν κάνω λάθο βγαίνουμε από το πακέτο, πια δεν είμαστε με στον προπολογισμό του 2006 και στο σημείο 12 τη ημερήσια διάταξη έχουμε ένα νέο στάδιο στην κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με το Ράιμερ Ευχαριστώ Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ σύντομα έχουμε μια πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την κινητοποίηση του Ταμείου παγκοσμιοποίηση, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Την έχουμε συζητήσει διεξοδικά. Έχουμε το μεταξύ και τη γνωμοδότηση Επιτροπή Απασχόληση. Την έχετε δει μέσα στα, κείμενα, στα έγγραφά σα, στο πρώτο τεύχο, με το λατινικό νούμερο 1. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι εν ώψη συζητήσεων τη τελευταία συνόδου Ολομελία στο Στρασβούργο, κατέστησα φες για το Ταμείο αυτό ότι δεν θα γίνεται η κινητοποίηση ταυτόχρονα για διάφορα ταμεία, για διάφορους τομείς μάλλον ε, και ότι θα γίνεται μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις έτσι ώστε να μπορούμε να κινούμαστε ταχύτερα και να δίνουμε περισσότερη έμφαση στα προβλήματα στα οποία εντοπίζουμε και να συζητούμε ενδεχομένω ε, ό,τι χρειάζεται. Και επίση και η Επιτροπή μας υπεσχέθη αντίστοιχη στάση. Γι' αυτό λοιπόν προσμένω στην κινητοποίηση αυτή με τις τρεις προτάσεις που βλέπουμε ε, να έχουμε την τελευταία πρόταση, την τελευταία φορά που μα ζητούν ταυτόχρονα να κινητοποιήσουμε το Ταμείο για τρεις περιπτώσεις μαζί. Ελπίζω να μας το επιβεβαιώσει και η Επιτροπή σήμερα. Είχαμε τις ερωτήσεις μας, τις διατυπώσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση, μαζί με τις ε, παρατηρήσεις όπως είπα και της Επιτροπής Απασχόλησης, όπου βλέπετε και κάποιες απαντήσεις από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Είναι οι περιπτώσεις, οι υποθέσεις μάλλον Volvo, με 1.500 εργαζομένους από τους 4.687 συνολικά απολυμμένους θα εξασφαλίσουν ε, οικονομική υποστήριξη. εφόσον πληρούνται βέβαια όλες οι προδιαγραφές, αν και χρειάζονται σε ορισμένα σημεία επιπλέον πληροφορίες ως προς εκείνους οι οποίοι έχουν λάβει την υποστήριξη, την ενίσχυση και τα νούμερα. Επίσης, το αίτημα το σχετικό με την Αυστρία, όπου καθίσατε σαφές ότι υπάρχουν διαφορετικά ποσά, προβλέπονται διαφορετικά ποσά ανά εργαζόμενο στους, ε, στην Σουηδία παραδείγματι είχαν στηθεί 6.500 ευρώ για κάθε εργαζόμενο, για την Αυστρία 14.300 ανά εργαζόμενο. Είναι μια συζήτηση που έχουμε ξανακάνει ούτως ή άλλως και η Επιτροπή είχε ε, δώσει κάποιες απαντήσεις. Εδώ την υπόθεση της επιχειρήσης Heymans στις κατοχώρες, Ιδιαίτερα με το σημείο 3 υπογραμμίζουμε την ανάγκη η χρηματοοικονομική ενίσχυση να μην αντικαταστήσει μέτρα που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων. Είναι συμπληρωματική αυτή η ενίσχυση μόνο. Και το άρθρο 12 4 του κανονισμού, σας το λέω άλλωστε στα αγγλικά, υπενθυμίζουμε στην Επιτροπή ότι απαιτεί και στοιχεία ικανοποιητικά ότι τα κριτήρια του άρθρου 2.6 έχουν τηρηθεί και ότι τα κράτη-μέλη ε, τα κράτη-μέλη δεν είναι ικανοποιημένοι από την απλή μάλλον οι βουλευτές δεν είναι ικανοποιημένοι από την απλή επιβεβαίωση ότι τα μέτρα αυτά θα είναι συμπληρωματικά. Θέλουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία δηλαδή. Και γι' αυτό, Πρόεδρε, για να συνεχίσω, θα ήθελα να δοθεί ευκαιρία και στην Επιτροπή να μα δώσει κάποιε απαντήσει πιο συγκεκριμένα, σύντομε, στι παρατηρήσει αυτέ. Ο Πρόεδρος. Θέλουν οι συνάδελφοι να συμπληρώσουν δεχομένως με άλλες ερωτήσεις προς την Επιτροπή, κύριος Φέρλαντς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Φερνάντς. Για το σημείο 12, αλλά και για το σημείο 13. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην ε, παγκοσμιοποίηση. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι ένα ταμείο το οποίο θα πρέπει να ε, στηρίξει εργαζομένους ή απολυμένους. Ενώ το διαρθρωτικό ταμείο έχει άλλο ρόλο, μακροπρόθεσμο, στο διαρθρωτικό, δεν είναι δηλαδή σε ε, σχέση ε, συμπληρωματικό, μάλλον δεν αντικαθιστά το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης, αλλά είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους, είναι παραπληρωματικά μεταξύ τους τα δύο ταμεία. Μπορούμε ενδεχομένως να αμφισβητήσουμε την αποτελεσματικότητα του Ταμείου που στόχος έχει να εξασφαλίσει την πλήρη απασχόληση και, ή τις διατυπώσεις απορρόφησης των κονδυλίων του, αξιοποίησης του, αφού βλέπουμε πόσο υψηλά είναι τα ποσοστά της ανεργίας. Αλλά, αλλά το κοινωνικό ταμείο, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που έχει διαρθρωτικό ρόλο, που εξυπηρετεί το στόχο της συνοχής και μακροπρόθεσμα ε, στοχεύει μόνο, δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο είναι ένα ταμείο για τη μετώπιση συγκεκριμένων και στιγμιαίων ουσιαστικά αναγκών. Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση λοιπόν δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από το ή εις βάρος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ευχαριστώ. κύριος Γκαρίγα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για αυτά που είπε ο συνάδελφος Φερνάντες, νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει κάποια αριθμητικά στοιχεία για το ποιες, ε, ποιο τμήμα των ποσοτήτων που κινητοποιήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ε, ήρθαν από προήρθαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Διότι εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι όλα αυτά τα οποία χρηματοδοτούμε τελευταίως από το Ταμείο προσαρμογή στην Πιαγκοσμιοποίηση προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και όπως είπε και ο συνάδελφο, αυτή δεν είναι αρχική πρόθεση του Ταμείου, ούτε αυτό που ψηφίσαμε εμεί το 2006. Θα ήθελα λοιπόν να μου δοθούν ε, τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ, Φέρ. Ε, η συζήτηση αυτή σχετίζεται στενά με αυτά που πρέπει να κάνουμε για το σημείο 13. Και για τη Γιούτα Χάουκ θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ πολύ με τα όσα είπε ο κύριος Φερνάντος και ο κύριος ε, Γαρίγκα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε πάντα όταν κάνουμε μεταφορές από το κοινωνικό τομείο αλλά δεν βρήκε άλλη εναλλακτική Γιούτα Χάουκ και γι' αυτό μας προτείνει να εγκρίνουμε την ε, μεταφορά αλλά με τι ίδιες επιφυλάξει και τα ίδια προβλήματα που επισήμαναν και οι κύριοι Φερνάνης και Γαρίγα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Αρκετέ είναι ερωτήσει προ την Επιτροπή. Έχουμε στου φακέλους μα. την γνωμοδότηση που αφορά την υπόθεση Volvo, την στηρία της Αυστρίας και την επιχείρηση Χάιμαν στο κατών χωρών. Υπάρχουν παρατηρήσει τη Επιτροπή Απασχόληση που είδατε, αλλά και οι συνάδελφοι έχουν διατυπώσει παρατηρήσει και ερωτήσει. Ρωτώ την Επιτροπή αν είσαι θέση να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την πρώτη. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι όντως ε, ε, θα γίνεται μεμονωμένα η προβολή των υποθέσεων, παρουσίαση των θεμάτων για ενίσχυση. Ίσως θα είναι και χρήσιμο να γίνει μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων, αν θέλετε, για να προσδιορίζουμε κάποιες βασικές προδιαγραφές, γιατί θα έχουμε αιτήματα για μεταφορές κονδυλίων που ε, θα έρχονται όλο και πιο συχνά, θα είναι όλο και πιο πυκνά και βέβαια αυτό θα επηρεάσει και τι διαδικασίε για τη λήψη αποφάσεων και το χρόνο που θα πρέπει να αφιερώνει η Επιτροπή σα ενδεχομένω στην έξοδο των θεμάτων αυτών. Και γι' αυτό θα θέλαμε να, ξεκινήσουμε μια διαδικασία άτυπη που θα διευκολύνει την ε, ανταλλαγή απόψεων και την διατύπωση των ε, προτάσεων ε, και φυσικά την έγκρισή τους. Τώρα, για τις σχέσεις του Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Αντιμετώπισης Παγκοσμιοποίησης. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι εις βάρος του Κοινωνικού Ταμείου, δηλαδή γιατί τα κονδύλια για το Ταμείο Αντιμετώπισης Παγκοσμιοποίησης προέρχεται από τι ε, αναλήψει υποχρεώσεων που έχουν εγγραφεί στον προπολογισμό από την αρχή του χρόνου εφόσον, προϋπο, πληρούνται οι προποθέσει από το ειδικό αποθεματικό δηλαδή που έχει προβλεφθεί για αυτό το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Οι μεταφορέ, όταν έχουν να κάνουν με πιστώσεις από το Κοινωνικό Ταμείο αφορούν πιστώσεις πληρωμών. Από πλευρά τη Επιτροπή, λοιπόν, εγώ θα μπορούσα να σα προτείνω να σα αποστείλουμε τις, ε, ε, τα ποσά που απορροφήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια που έχει δραστηριοποιηθεί το ταμείο αυτό και να σας εξηγήσω τα ποσοστά ε, επί του συνόλου των πιστώσεων πληρωμών του Κοινωνικού Ταμείου ότι είναι μόνο 1% και επίσης θα μπορούσα να σας δώσω και ποσοστά αξιοποίηση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τα τρία τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και του 2009. Με ένα επίπεδο αξιοποίηση αυτών των ε, πιστώσεων πληρωμών χαμηλό τερό κατάτι από το 100%. Σχεδόν 100% λοιπόν. Άρα η αξιοποίηση των ε, πιστώσεων πληρωμών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δεν ε, αποβαίνει εις βάρος του μέσου του ίδιου. Δεν έχει επηρεαστεί δηλαδή η εφαρμογή του προγράμματος αυτού από την ε, απορρόφηση κάποιων μικρών κονδύλων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Για δε τις διαβεβαιώσεις που προσφέρουν τα κράτη-μέλη για τα μέτρα τα οποία προβλέπονται από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που δεν έχουν καλυφθεί από άλλα δημοσιονομικά μέσα ή εργαλεία, όργανα. Ε, ασφαλώς εδώ νομίζω ότι αυτό ζήτημα αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία πρέπει να αποτελεί και τη βάση τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Εφόσον χρειαστεί μπορούμε να συζητήσουμε σε λεπτομέρειε το θέμα αυτό. Αλλά ω εκκίνηση, ω σημείο αφετηρία, πιστεύω, πρέπει να έχουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Για τον τρόπο με τον οποίο να αξιοποιείται το μέσο. Ευχαριστώ κύριο Κουτμάνος. Για το 12 και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω λίγο αργότερα και στο 15 στην ημερήσια διάταξη. Αυτό που βλέπω εγώ σε επικίνδυνο είναι ότι αν συνεχίσει το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και δεν προβλέπεται, συγκεκριμένη γραμμή στον προπολογισμό για τι ε, δαπάνε του, αργά ή γρήγορα θα απορροφήσει χρήματα από το, ταμείο, από το ε, κοινωνικό ταμείο. Όντως, 500 εκατομμύρια συνολικό ποσό, εάν όλη η γραμμή εξαντληθεί, θα αποδειχθεί ότι είναι περιορισμένο ποσό, εάν ε, κοιτάξουμε τα μη απορροπηθέντα ποσά από τις πληρωμές των διαρθρωτικών ταμείων. Ναι, αλλά τα ποσά των διαρθρωτικών ταμείων μεταφέρονται, γίνονται rollover. Εάν δούμε δηλαδή από το 2006 ποσά υπάρχουν ακόμη 16 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα που δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί. Άρα, θα πρέπει να δούμε πότε θα ζητούνται τα χρήματα και μέχρι την ώρα που θα ζητούν τα χρήματα αυτά από το κοινωνικό ταμείο, Όντω μπορούν από εκεί να, ε, να βγαίνουν χρήματα για το παγκοσμιοποίηση εφόσον κάποια κράτη δεν ε, τα διεκδικούν. Και ίσως για το 2006 μπορεί να μην έχουμε 95% αλλά 85-86% πληρωμές για ορισμένα κράτη τα οποία χάνουν την ευκαιρία τους και έτσι τα χρήματα μπορούν να πηγαίνουν στη συγκεκριμένη αυτή ανάγκη. Το θέμα όμω είναι ότι εάν βελτιώσουν την ικανότητα απορρόφησης, μάλλον την πειθαρχία του στα κράτη, το προ το πειθαρχία τους, τότε δεν θα περισσεύουν αυτά τα λεφτά. θα μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιούμε για το Ταμείο παγκοσμιοποίηση, κονδύλια του, ταμείου, του Κοινωνικού Ταμείου. Εάν η ποιοτική προσέγγιση για τις ε, πληρωμές του, για την κινητοποίηση του Ταμείου ε, βελτιωθούν, τότε δεν θα μπορούμε καν να το χρησιμοποιήσουμε. Γιατί διαφορετικά δεν προβλέπονται άλλοι πόροι για το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Από, το, από τα διευθυντικά ταμεία μόνο παίρνουμε κονδύλια τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί για λόγου ε, μη ικανοποίηση, μη ε, επιτέλεση των υποχρεώσεων από πλευρά των κρατών μέλων. Τα κράτη-μέλη δηλαδή έχουν κάπου ε, υστερήσει ω προ τι υποχρεώσει του και τότε ε, μπορούν να διατεθούν τα, τα, χρήματα αυτά στο Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Αν όμω βελτιώσουν τι επιδόσει στα κράτη-μέλη και πάνω απ' όλα, το, μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή να διαθέσουμε τα κονδύλια. Ενώ θα χρειαζόμαστε όλο και περισσότερη στήριξη. Τι θα γίνει, δηλαδή, εδώ έχουμε να κάνουμε μια φιλοσοφική, με ένα φιλοσοφικό πρόβλημα. Τι θα κάνουμε όταν σιγά-σιγά έχουμε όλο και περισσότερε ανάγκε στο Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφοι, πολύ εύστοχη παρατήρηση. χρηματοδότηση από το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση μπορούμε να προβλέψουμε μόνο στο βαθμό που οι πιστώσει ε, που έχουν διατεθεί στα διαφορετικά ταμεία δεν εξατλούνται. Με τον ίδιο τρόπο που έγινε η χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια κάποιων έκτακτων και τελείως διαφορετικής φύσεως δαπανών και, από, και το Γαλιλαίο και το Recovery Plan και το Milk Fund, το Ταμείο Γάλακτος γιατί, διότι υπήρξαν κάποια ποσά ε, που είχαν αγραφεί στο προπολογισμό στη δεύτερη κατηγορία, στο στον γεωργικό προπολογισμό, αλλά δεν απορροφήθηκαν. Κύριε Σιγητά, ακούσατε τις παρατηρήσεις των συναδέλφων, ακούσατε και τις απαντήσεις Επιτροπής. Πού καταλήγετε. Λοιπόν, καταρχάς δεν θέλω να σταματήσω την κινητοποίηση του Ταμείου σε αυτές τις περιπτώσεις. Θέλω να συστήσω στην Επιτροπή την υπερψήφιση. Ακόμα τότε τη βδομάδα θα συναντηθώ με την ειδική ομάδα που έχει συσταθεί από την Επιτροπή Απασχόλησης ε, και ασχολείται με το θέμα και καλά κάνει και θα αξιολογήσουμε, θα αναθεωρήσουμε το ταμείο αυτό έχοντας υπόψη όλα αυτά τα θέματα και η σχέση με το κοινωνικό ταμείο και η χρηματοδότηση πώς έχει. Θα δούμε και πώς ε, μπορεί να μεταφέρεται ένα τέτοιο ταμείο ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Όλα αυτά εκκρεμούν και θα τα συζητήσουμε ζητήματα. Και πριν από λίγους μήνες διευκολύναμε την πρόσβαση στο ταμείο αυτό, διότι διαπιστώσαμε ότι τα χρήματα που θεωρητικά υπάρχουν, μας το είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, υποαπορροφούνται και δεν έχουν σε κανένα βαθμό εξαντληθεί. Τώρα επιταχύνονται οι διαδικασίες και ανεξάρτητα τώρα από το κοινωνικό ταμείο ή από τα διορθωτικά ταμεία, γενικά τα περιθώρια τα επόμενα έτη σε όλες τις κατηγορίες του προϋπολογισμού στενεύουν, για να μην πω ότι στερεύουν κιόλα. Και ε, θα πρέπει να το δούμε όλο αυτό το θέμα σε μια νέα δυναμική και μπορούμε. Για σήμερα όμως σας συνιστώ να υπερψηφίσουμε ε, αυτό το θέμα και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης να χαράξουμε στρατηγική για τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ ο Πρόεδρος. Οπότε, θα υποβάλω τώρα αυτό ε, σε ψήφιση και είναι τελευταία φορά που μία μόνο ψηφοφορία ισχύει για πολλές ταυτόχρονα δράσεις ε, και χρηματοδοτήσεις. Επιμείναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταρχήν συμφώνησε στο εξή η νομική βάση να είναι όπως για τις πιστώσεις εξειδικευμένη ανά ε, κονδύλι και ανά δράση για να αποφύγουμε την κατάσταση που γνωρίσαμε πριν από λίγες εβδομάδες όταν είχαμε λάβει μία απόφαση για δύο ε, δράσεις που δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους και δεν είχαμε την ίδια αντίδραση εμείς. Στη, στο Βέλιο και στην Ιρλανδία ήταν οι δύο περιπτώσεις. Λοιπόν, ε, ποιος είναι υπέρ της απόφασης αυτής που προτείνει ο συγητής μας. Ευχαριστώ. Κατά. Μία ψήφος κατά και αποχές δεν έχουμε. Καλώς. Ε, ούτως αποφασίζεται. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σίτη και παίρνουμε στο σημείο 13 συνεπώς απουσία της Γιούτα Χάουκ Ευχαριστώ τον Γεράν Χέρν που αναλαμβάνει να ε, είναι αναπληρωτής συζήτη και το δέχεται. Η πρώτη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων είναι το 48 που μόλις ψηφίσαμε. Εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είναι υπέρ, ψήφι υπέρ της μεταφοράς αυτής. Οι ίδιοι υποθέτω. Ευχαριστώ κατά. Οι ίδιοι αποχές Εγκρίνεται η μεταφορά υπαριθμών 48. Έχει και άλλη μεταφορά πιστώσεων, 58, 56, συγγνώμη. Ναι, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Πρόκειται για μια μεταφορά που αφορά συμπληρωματικέ δαπάνε. Δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσό αλλά αυτέ είναι αναλήψεις υποχρεώσεων που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα. Επομένω, είμαστε υπέρ. Το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να το καθυστερήσουμε, αλλά η Γιούτα Χάουκ προτείνει να το υπερψηφίσουμε. Σα ευχαριστώ. Δεν θέλει κανεί το λόγο. Ψήφι υπέρ ε, της μεταφοράς που προτείνει ο εισηγητή μα. Ε, κατά, ε, μία ψήφο ε, κατά, αποχέ. χωρίς αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν και η μεταφορά αυτή. Δεν έχουμε άλλες αιτήσει μεταφοράς πιστώσεων για τον κύριο Φέρμ και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 14, λοιπά τμήματα. Η συγκητή εδώ είναι ο κύριος Λεβαντόφσκι και έχει μια μεταφορά πίστος για το κοινοβούλιο που λέγεται C22. Κύριε συγκητά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρωινή μας συνεδρίαση είχε πολλές συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ τώρα είμαστε στα λοιπά όργανα. Συζητάμε το θέμα της αγοράς του κτηρίου της ε, οδού Τρεύ. Με έπεισαν ο κύριος ε, Βιντάλ Κουάντρα και ο Σελβατόρ ε, Γκαρίγκα Πογέδου για το θέμα αυτό και υπήρξε και μια επιστολή του Προέδρου μας, ε, του κυρίου Λαμασούρ, προς το Προεδρείο. Έχουμε απάντηση για το θέμα του αμοιάντου. Και για το Τρεβένα θεωρούμε ότι έχει ε, υπάρξει αναλογικότητα. Τώρα θα πρέπει να δούμε πρώτα το C24. Το C24 επαναλαμβάνω, διότι αυτό αφορά τις άλλες αγορές, οι οποίες θα πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής για τα κτίρια, διότι το C24 αφορά το τι θα γίνει μετά όσα παραμένουν από το αποθεματικό για τα κτίρια. Αυτή είναι Συγγνώμη, διακόπτει ο Πρόεδρος. Συγγνώμη, κύριε Σίγητα. Σας προτείνω προς το παρόν να αφήσουμε τη μεταφορά υπαριθμών 24 που αφορά ε, το κτίριο που θα αγοράσουμε ενδεχομένω στη Βουδαπέστη. να ε, ε, το αφήσουμε αυτό στην άκρη προς στιγμή, διότι πρώτα θα πρέπει να εξετάσουμε επί της ουσίας το θέμα στην έκθεση της κυρίας Χολμάγερ και είναι το επόμενο σημείο. Και από την άλλη, καλέσαμε τον αρμόδιο αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, αρμόδιο για τα κτίρια που είναι ο κύριος Βιντάλ Κουάδρας και θα έρθει σε δεκάμιση. Αν δεν σας πειράζει, θα προτιμούσα να δούμε πρώτα τις άλλες μεταφορές πιστώσεων και να αφήσουμε αυτό στην άκρη. Εσείς είστε η αρχή εδώ, ο αρχηγός της Επιτροπής. Ωραία, να δούμε το C22. Αυτό και πάλι αφορά εφαρμογή απόφαση του Προεδρείου, που ενισχύει την εξωτερική βοήθεια στον τομέα του συστήματος λογισμικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 2009 στον προπολογισμό είχαμε διαθέσει περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή τη γραμμή προπολογισμού για το θέμα αυτό και θα έρουμε ενίσχυση ενός εκατομμυρίου 150.000 ευρώ, α, συγγνώμη, ενός 850.000 ευρώ. Αυτό ε, κατέληξε ως συμπέρασμα του εξωτερικού ελέγχου για τα τμήματα υπολογιστών του Λουξεμβούργου και των Βρυξελών εκτός του κτίριου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μην υπάρχουν προβλήματα με την ε, ηλεκτροδότηση Κατ' εμέ λοιπόν είναι δικαιολογημένο, διότι ήταν αποτέλεσμα της απόφασης του εξωτερικού ελέγχου. Τα υπόλοιπα είναι για να γίνουν δύο μελέτες. Η μελέτη EMAS και ε, μία μελέτη για την κάλυψη με Wi-Fi. Ε, και οι δύο στοιχίζουν από 250.000 ευρώ και δεν θα πρέπει να έχουμε καμία ένσταση, διότι υπάρχει αποθεματικό ε, στο θέμα των της επίπλωσης και του λογισμικού, επομένως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά. Ε, δεν είναι δώρο Χριστουγέννων αυτές οι μεταφορές, αλλά είμαι θετικός. Κυρίως ε, λόγω της αιτιολόγησης που δόθηκε για αυτές τις μεταφορές. Θέλουμε να ενισχύσουμε το λογισμικό του Κοινοβουλίου και εγώ δεν ρώτησα λεπτομέρειες ε, για τα θέματα αυτά, γιατί είμαι τη εποχή προ προ-υπολογιστών. Εκ δεξιών και εξ αριστερών έχω τη νέα γενιά, μπορείτε να ρωτήσετε αυτούς. Καλώ ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Πάντως μπορούμε εδώ να διαπιστώσουμε ότι το Προεδρείο χρησιμοποίησε καλά την προηγούμενη μεταφορά που μας είχε προτείνει ο κύριος Λεβαντόφσκι, γιατί επιτέλους μπορούμε να πλύνουμε τα χέρια μας. Ο κύριος Λεβαντόφσκι είχε προτείνει να απελευθερώσουμε χρήματα για είδη καθαριότητας, αλλά όχι για υπηρεσίες. Και έχουμε σε ώρα τα έδρανα ε, μαντιλάκια ε, για απολύμανση και ο καθένας που μιλάει <laughs> μετά νύπτει τα σχήρες του με ένα τέτοιο πολυμαντικό μαντιλάκι. Λοιπόν, ε, ο Βαλάντι Μάνκα έχει ζητήσει το λόγο πριν ψηφίσουμε, που είναι ο εισηγητή για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου και θέλει να πει τη γνώμη του. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ, αλλά έχω μια ερώτηση. Εδώ έχω ένα υπολογιστή και πάντα χρησιμοποιώ ασύρματο ε, διαδίκτυο. Και είμαι πολύ ικανοποιημένο γιατί το, έχουμε σε όλε τι αίθουσε συνεδριάσεων. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εφαρμογή. Τώρα θέλουμε να αναθέσουμε μελέτη για το Wi-Fi, ε, για να έχουμε ε, ασύρματο ε, διαδίκτυο και στους διαδρόμους. Γιατί να δώσουμε 250.000 ευρώ. Για ποιο λόγο. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε και στο διάδρομο ασύρματο ίντερνετ. Δεν μας στάνει στις αίθουσες. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος στην πρόσβαση που έχουμε στο δίκτυο όπως έχει αυτή τη στιγμή. Γιατί, ε, ρωτώ, για ποιο λόγο να θέσουμε τέτοια μελέτη. Ευχαριστώ πολύ, καλώς. Ο αρμόδιος γενικός διευθυντής είναι παρόν και θα απαντήσει σίγουρα στην ερώτηση αυτή. Έχω όμως και μια άλλη ερώτηση από τον κύριο Χάγλοντ που ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με αυτά που μόλις είπε ο κύριος Μάνκα, εγώ είμαι από αυτού τη νέα γενιά που πιστεύουν ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει να μα διατίθεται παντού, όπως και το ηλεκτρικό ρεύμα. Χαίρομαι λοιπόν που ε, αλλάζει η κατάσταση εδώ. Η κατάσταση δημιουργεί προβλήματα σε κάποιους που ούτως ή άλλως είναι συνηθισμένοι να χρησιμοποιουν WIFI. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρειαζόμαστε μελέτη. Μπορούμε απλά να διαθέσουμε τα κονδύλια αυτά για να εξοπλίσουμε όλα μας τα κτίρια με ασύρματη σύνδεση. Εμείς ε, από πλευράς πολιτικών ομάδας θα θέλαμε να προχωρήσει το θέμα αυτό όσο το δυνατό γρηγορότερα και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λεβαντόφσκι αν θέλετε να συμπεριλάβετε και τις πολιτικές ομάδες ε, στην ε, υλοποίηση. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κύριος Γενικός Διευθυντής επιθυμεί να μιλήσει για να δώσει κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μάλιστα μερικές διευκρινήσεις. Αποφάσισε το Προεδρείο να αναθέσουμε γενική μελέτη για την επέκταση του ασυρμάτου δικτύου. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα μέτρα που αφορά η μελέτη, ανακτήριο. Περιοριζόμαστε όμως στα κοινοβουλευτικά κτίρια για να δούμε πού μπορούμε να βάλουμε κεραίες για να καλύπτουν τον απαραίτητο χώρο χωρίς να είναι υπερβολική η κάλυψη. Ε, στα δύο ημικύκλια επίσης ε, έχει ζητηθεί και στι Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο να υπάρχει κάλυψη με ασύρματο γιατί προς στιγμή δεν έχει αποφασίσει το Προεδρείο για το ασύρματο διαδίκτυο στην Ολομέλεια. Υπάρχουν όμω αιτήματα και βεβαίω οι βουλευτές που θέλουν να συμμετέχουν στι μελέτε μπορούν να συμμετέχουν, να συμπεριληφθούν στην εργασία αυτή. Ευχαριστώ. Σας επιβεβαίωνω ότι οι πολιτικές ομάδες βεβαίως θέλουν να συμμετέχουν στη μελέτη αυτή. Υποθέτω ότι εδώ σας δίνω την αίσθηση όλων των πολιτικών ομάδων. Και συμφωνώ και εγώ με τη νέα ε, γενιά ότι χρειαζόμαστε παντού ασύρματο διαδίκτυο και στην Ολομέλεια να έχουμε κάλυψη. Κύριε τι προτείνετε λοιπόν μετά από όλα αυτά που ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ξέχασα να σας το πω, αλλά σαφώς θα πρέπει να εποπτεύουμε τα αποτελέσματα της μελέτης και οι πολιτικές ομάδες σαφώς πρέπει να συμμετέχουν στην εφαρμογή. Αυτό είναι σαφές για μένα. Επομένως, η σύστασή μου είναι θετική, αφού ακούσαμε και τις ε, επεξηγήσεις. Ευχαριστώ. Ποιος είναι λοιπόν υπέρ αυτής της μεταφοράς πιστώσεων, υπέρ 22, που μας προτείνει ο συγητής μας, με τις προφορικές παρατηρήσεις που ακολούθησαν. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Δύο κατά. Αποχές. Η σοσιαλιστική ομάδα απέχει. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται τη μεταφορά πιστώσα. Τώρα ερχόμαστε στο σχέδιο μεταφοράς πιστώσεων της Επιτροπής Περιφερειών. Κύριε Σιγητά μου. Προτάσει από την Επιτροπή Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα πρέπει να συζητηθούν από κοινού, διότι είναι το ίδιο θέμα αντικατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αποσύρθηκε το 1 τέταρτο των υπολογιστών και εδώ έχουμε τα υπόλοιπα τη συζήτηση για τη μεταφορά που είχαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Είχαμε διαχωρίσει το θέμα των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τις άλλες ε, μεταφορές για την Επιτροπή των Περιφερειών και την ΟΚΕ. Και τώρα έχουμε κάποιες επιπλέον εξηγήσει. Δεν μπορώ να συμφωνήσω πλήρως με τις επεξηγήσει της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία ισχυρίζεται ότι το 2010 έχει μικρότερη ανάθεση κονδυλίων από ότι το 2009. Υπήρξε σχετική τροπολογία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ποσό για την επεξεργασία δεδομένων ε, συντήρηση και αγορά εξοπλισμού είναι υψηλότερο από ότι το 2009. Το επιχείρημά τους βέβαια είναι κάπως πιστικό, διότι και τα δύο όργανα συνεισέφεραν σε αποταμίευση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στην ε, συνδιαλλαγή και αυτό διευκόλυνε και τη συμφωνία και αυτό ήταν ε, τμήμα του θαύματος που είχαμε στον τίτλο 5 για τη ε, διαδικασία της συνδιαλλαγής. Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν να δώσουμε το πράσινο φως για να προχωρήσουμε στους υπολογιστέ, διότι το συνολικό ποσό το οποίο από τα εξοικονομήσαμε είναι πολύ πολύ ψηλότερο. Και αυτό που ζητά η Επιτροπή των Περιφερειών είναι 300.000 ευρώ και η ΕΟΚΕ 50.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα επιπλέον επιχείρημα λοιπόν για να συνεχίσει αυτό το σκεπτικό ανανέωσης του εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και στα δύο όργανα. Μας βοήθησαν να καταλήξουμε σε συμφωνία ε, στη διάρκεια της συνδιαλλαγής. Merci, Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Οπότε Άρα λέμε στα δύο αυτά θεσμικά όργανα ότι σας πήραμε χρήματα για να βρούμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο και τώρα σας επιτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε τα ολίγα που σας έχουμε αφήσει και να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Ακόμα και αν δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι θα πιάσουν τόπο. Εν πάση περιπτώσει κάπου ε, αυτό είναι. Και θα χαρούν οι νέοι γιατί τα χρήματα αυτά θα πάνε στην αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων εργαλείων πληροφορική τελευταίας τεχνολογίας. Δεν θέλει κανεί το λόγο από αυτού. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν και τις δύο μεταφορές πιστώσεων ε, ταυτόχρονα, γιατί πρόκειται για δύο όργανα αλλά για το ίδιο θέμα. Ευχαριστώ. Υπέρ. Κατά. Με τρεις ψήφους κατά. Ε, αποχές έχουμε. Όχι. Οπότε, η ΔΕΚ 1 και ΔΕΚ 2, οι μεταφορές πιστώσεων για την Επιτροπή Περιφερειών και την ΟΚΕ, εγκρίνονται. Τούτων εχθέντων, α, με την επιφύλαξη πάντα της 24, στην οποία θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, ερχόμαστε στο σημείο 15, εφαρμογή της πολιτικής συνοχής Ο κύριος Γκοντμάνης θα μας παρουσιάσει το θέμα αυτό και την κατάσταση ως προς το θέμα και μετά από την πρόταση της Εκθέσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύντομη ανταλλαγή απόψεων ακολουθεί. Έχετε το λόγο αγαπητέ μου, κύριε Γκοτμάνης. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν είναι εύκολη η δουλειά μου. Είμαι ένα πληρωματικό μέλο στην Επιτροπή των Περιφερειών και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Ε, πάντα, δεν, πάντα έχουμε πρόβλημα με τα κονδύλια, δεν αρκούν τα χρήματα, δύσκολες διαδικασίε, δύσκολο να τηρηθούν. Εάν πρέπει να δούμε από την έποψη των προϋπολογισμών την υπόθεση αυτή, όμως βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα. Να σας δώσω κάποιες βασικές ιδέες, λοιπόν. Με βάση, τον, ε, με βάση την πίστοση 1083 θα διατεθούν τα κονδύλια αυτά και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να διαβάσουμε και τον κανονισμό. Το 2009, εφέτος τον Απρίλιο δηλαδή, τροποποιήθηκε ο κανονισμός κατά ένα πράγμα από την Επιτροπή, την αύξηση των προκαταβολών. Δηλαδή, οι πληρωμέ από την Επιτροπή, οι προκαταβολέ μάλλον από την Επιτροπή, αυξάνονται, ενισχύονται για το περιφερειακό και, τα, και το κοινωνικό ταμείο. Από 2 σε 3%. Όχι όμω το Ταμείο συνοχή. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε ότι βελτιώνεται η κατάσταση για τι χώρε που παίρνουν χρήματα. Όμω, από την έπαψη των προπολογισμών υπάρχει εξή δυσκολία. Ότι αν ξεχωρίσουμε το παρελθόν από το μέλλον και το παρόν φυσικά, τι κάνουμε, έχουμε ως παρελθόν το 2000 με 2006, την περίοδο 2000-2006. Διαθέτουμε χρήματα στα κράτη-μέλη επί τη βάση της ε, επιστροφής, του rollover, της μετακύλησης δηλαδή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για δύο ταμεία, το κοινωνικό και το ε, περιφερειακό, έκλεισε πλέον η προθεσμία, γιατί ήταν η 1η Ιανουαρίου του 2009. Αν λοιπόν η σχετική τεκμήριο στα απαραίτητα έγγραφα δεν μπόρεσαν να κατευθούν εγκαίρως στην Επιτροπή, τυπικά δεν υπευλίζαν στην Επιτροπή, τα χάσαν τα λεφτά τα κράτη-μέλη. Επισήμως. Επισήμως. Πρέπει λοιπόν να ρωτήσω από την Επιτροπή να, με, να μου επιβεβαιώσει αν όντω αυτό ισχύει ή αν υπάρχει ένα περιθώριο μεγαλύτερο για τι χώρε, οι οποίε δεν τήρησαν τι προθεσμίε. Διότι αν υπάρχει ένα περιθώριο, τότε πρέπει να υπολογίσουμε και τα επιπλέον κονδύλια που θα πρέπει να τεθούν. Και εδώ έχουμε να κάνουμε 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλα τα, τα ποσά, δεν είναι ψίχουλα. Για το Ταμείο συνοχή, όμω τα πράγματα είναι διαφορετικά, διότι η προθεσμία του Ταμείου Συνοχή ήταν 31 Δεκεμβρίου του 2010. Άρα υπάρχει ακόμη περιθώριο και είναι μεγάλο διάστημα από το 2006 μέχρι τώρα. Τέσσερα χρόνια. Και ακόμη μπορεί η Επιτροπή επί τη βάση της απόδοσης του, ε, του reimbursement να ζητήσει τα κονδύλια αυτά. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί αν δούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν και τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, υπάρχουν χώρε οι οποίε δεν έχουν εκπληρώσει τι υποχρεώσει του, χωρί να θέλω να τι αναφέρω ονομαστικά. Αλλά είναι η πρώτη φορά που έχω δει κάποιε πληροφορίε συγκεκριμένε και πρέπει να τι κοιτάξω πολύ προσεκτικά και διαπιστώνω σε σχέση με το παρελθόν ότι 95% το, το ποσοστό της επιστροφής, δηλαδή τα ποσά τα οποία είναι κατανεμημένα σε δεσμεύσεις, 95% που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλονται και 5% μένουν στο αποθεματικό και καταβάλλονται αργότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα ως μέλος. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, είχαν κάποιες χώρες 88%, 86%, 8 με 10% δηλαδή κάτω από το απαραίτητο ποσοστό που απαιτείται για να ε, έχει εκπληρώσει το κράτος στο σύνολο της υποχρεώσεις του. Για το κοινωνικό ταμείο, κάποιες χώρες είναι μέχρι το 73% μόνο, δηλαδή έχουν απόκληση ε, μέχρι και 22% από το ποσοστό που θα έπρεπε να έχουν επιτύχει. Άρα, το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα γίνει με το ποσό αυτό που ε, περισσεύει, το εκκρεμές αυτό ποσό. Ή θα πρέπει να καταβληθεί βάσει του προγράμματος του σχεδίου συνοχής, όπου θα πρέπει τα ε, στοιχεία να παρουσιαστούν μέχρι τα 31 Δεκεμβρίου του 2010, ή θα πρέπει να εγκρίνει η Επιτροπή μας αυτό το ποσό, επιπλέον, που θα προτείνει η Επιτροπή, ως επιπλέον ποσό για το Ταμείο για το Ταμείο Συνοχής. Και δεν μιλάω για το κοινωνικό ταμείο, το ανέφερα νωρίτερα γιατί σχετίζεται με την παγκοσμιοποίηση. Αλλά αν δούμε το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που ε, σε μεγάλο βαθμό ε, ενδιαφέρει τα κράτη-μέλη, για το 2000-2006 βλέπουμε πως υπάρχουν ε, χώρες με ποσοστό εκτέλεσης αντί για 95-85-86% και είμαι 87% το πολύ. Και όταν επιπλέον έρχεται η Επιτροπή για να στήσει με μια, επιπλέ... με μια νέα πρωτοβουλία, την πρωτοβουλία Urban και ξέρουν πολύ τι σημαίνει αυτό, σημαίνει δηλαδή ότι αγωνίστηκαν στι διάφορε χώρε ε, μέλη, οι πόλει, τα αστικά κέντρα δηλαδή για να διεκδικήσουν ένα ποσό από τη χρηματοδότηση, το ξέρω και από τη δική μου την πατρίδα, εκεί η εκτέλεση ήταν ακόμα χειρότερη από ό,τι στο παρελθόν, από ό,τι στα υπόλοιπα μάλλον κεφάλαια, 80, το πολύ πολύ 82% για ορισμένε περιπτώσει. Άρα δεν υπάρχει αρκετά καλή εκτέλεση των κοινωνικών ταμείων. Και το θέμα δεν είναι αν θα καθυστερήσουμε στις διαδικασίες και όλα αυτά. Όχι. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει πρόβλημα στην απορρόφηση, στην εκτέλεση και άρα τι θα κάνουμε. Το Ταμείο Αλίας επίσης που δεν είναι μεγάλο ταμείο. Αντί για 95% εκτέλεση έχουμε 1,83, 1,76% σε ορισμένες περιπτώσεις. Άρα Υπάρχουν χώρε οι οποίε στο παρελθόν δεν έχουν εκτελέσει τι επιτελέσει επιτροποχρώσεω και για μα από έποψη δημοσιονομική τίθεται το δίλημα. Δεν θα δώσουμε πια τίποτα, δεν θα διαθέσουμε τα κονδύλια αυτά πια που είναι στο αποθεματικό. Θα τα διαθέσουμε αργότερα, θα παραμείνουν κάπου, θα δεσμευτούμε για το μέλλον, θα εκτελεστεί η υποχρέωση της ανάκτησης των κονδυλίων που δεν έχουν εκτελεστεί. Μεγάλο πρόβλημα. Και για να δούμε και την ε, κατάσταση που έχουμε τώρα, την επίκαιρη κατάσταση, θα είδατε ίσως και από τις πληροφορίες από το Κόμπου News, δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Αυτό που πρέπει να κάνει μια χώρα για να εξασφαλίσει τα χρήματα αυτά θα είναι πρώτον να εγκρίνει ένα πλαίσιο, το μεγάλο πρόγραμμα, πράγμα που έχουν κάνει όλες οι χώρες. Το μεγάλο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεύτερον, να ε, εγκρίνει, να προσδιορίσει, να ορίσει ε, συστήματα ελέγχου της διαχείρισης που υπάρχουν και είναι καλά και θα δουν όλοι ότι ίσως προς το τέλος του χρόνου να έχει επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο. Όμως είμαστε στο 2009, το δε πρόβλημα ξεκινάει από το 2009, έστω δύο χρόνια, το 7, το 8 και το 9 μαζί, τρία χρόνια να το υπολογίσω, για να προβληθεί αυτό το, να προβληθεί αυτό το σχέδιο. Όμως αυτή είναι η μόνο τυπική προσέγγιση, γιατί μετά πρέπει να περάσουμε στα μεγάλα σχέδια, big projects, θα το δείτε και από τις εφημερίδες. 989 μεγάλα σχέδια που καλύπτουν όλες τις χώρες, όλα τα λειτουργικά προγράμματα. Από αυτά τα 989 Μόνο τα 150 τώρα έχουν διατεθεί στην Επιτροπή και μόνο έχουν κατατεθεί μάλλον στην Επιτροπή και μόνο 45 έχουν εγκριθεί. Πολύ χαμηλό το ποσοστό δηλαδή, μερικέ φορέ 4,5%. Και αν δεν έχει εγκριθεί το σχέδιο, το project, δεν μπορούν να διατεθούν και τα χρήματα. Το θέμα είναι ότι τα κράτη δεν είναι υποχρεωμένα να διατηρήσουν τον αριθμό των 989. Μπορεί να πάνε σε πιο μικρό αριθμό σχεδίων. Αλλά ε, μετά το θέμα πόσα σχέδια, πόσα project θα εγκρίνει η Επιτροπή, όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ότι με το σύστημα ελέγχου διαχείρισης, Management Control System. Αλλά το ζωοδέστατο είναι τα χρήματα που καταβάλλονται για ε, τα τεκμηρία, για τα έγγραφα, τα στοιχεία δηλαδή που διαθέτουν τα κράτη-μέλη. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι για όλα τα ταμεία, κατά μέσο όρο, φτάνουμε σε ποσοστό πληρωμών κατά 20% περίπου. Χρήματα, τα οποία δίνονται με βάση τα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή. Για όλα τα ταμεία όμω, υπάρχουν ποσοστά για ορισμένε χώρες. 40% για συνολικά για όλα τα ταμεία. 50, 41, 47% μεγάλη απόκληση λοιπόν. Και καθώς κάθε χώρα απαιτείται να, να καταθέσει δήλωση το 2009, το τέλος, το τέλος του 2009, για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν, εφαρμόστηκαν, εκτελέστηκαν τα κονδύλια αυτά. Και τα στοιχεία αυτά θα τα συλλέξει η Επιτροπή τον Απρίλιο του χρόνου για να δούμε συνολικά τι εικόνα παρουσιάζεται. Ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη εισρωή την τελευταία στιγμή στο παραπέντε, μέχρι το τέλος του χρόνου δηλαδή, ε, τεκμηρίων και ε, εγγράφων που χρειάζονται ε, και αντίστοιχα απαιτήσει για καταβολή των ποσών. Ερώτηση. Είμαστε έτοιμοι να ε, προσαρμοστούμε σε αυτή την επιταχυμένη διαδικασία και στη χαρτοπλημμύρα που θα προηγηθεί. Και δεν, αν αφήσουμε την ε, συνολική εικόνα των ταμείων και κοιτάξουμε χωριστά για το κάθε ταμείο, υπάρχουν χώρες που έχουν 49% για το διαστροτικό και άλλα για το κοινωνικό ταμείο και άλλα που έχουν 13 με πολύ μεγάλη, δηλαδή ένα προς τρία σχέση. Και για το, ταμείο, ε, για το περιφερειακό ταμείο υπάρχουν χώρες που έχουν ποσοστό 56% στις ε, πληρωμές. 4,5 δις που έχουν καταβληθεί από την αρχή ε, των προοπτικών. 4,5 όμως τι σημαίνει, ξέρετε. Τίποτα δεν είναι, ψίχουλα είναι. Διότι συνολικά το ποσό, το τελικό ποσό θα είναι 200 δις. Ψίχουλα λοιπόν το 4,5. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει, ε, το κρίσιμο ερώτημα θα είναι αν η ταχύτητα, ο ρυθμός δηλαδή που θα διατηρηθεί και αν θα μπορέσουμε, αν θα είναι χώρες που θα πάνε ε, με τον ε, κανόνα του νησιν 2, δύο χρόνια αργότερα δηλαδή, άλλες που θα κρατήσουν άλλους ρυθμούς. Και όσε δεν μπορούν να διατηρήσουν του υψηλού ρυθμού εκτέλεση θα χάσουν τα χρήματα αυτά. Για μερικέ χώρε μάλιστα είναι 900 εκατομμύρια ευρώ τα ποσά που θα χάσουν ξαφνικά. Για να μην μιλήσω για τα ταμεία συνοχή που είναι ακόμη τα πιο σοβαρά κονδύλια, τα πιο μεγάλα κονδύλια, όπου έχουμε χώρε με ποσοστό πληρωμών 9% ενώ άλλε έχουν 60% ποσοστό. Τεράστιες αποκλήσεις. Άρα, μεγάλο πρόβλημα και τα προβλήματα που μας επισημαίνει η Επιτροπή τα, κατανομή, τα κατανέμει σε τρεις ε, ομάδες. Υπάρχουν κάποιες χώρες για τις οποίες δεν προβλέπεται η δυνατότητα βελτίωσης του συστήματος ε, ελέγχου της διαχείρισης. Οπότε δεν μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο αυτές οι χώρες αυτές. Τελείωσε η ιστορία για αυτές, αν δεν βελτιώνεται αυτό το σύστημα. Άρα ερώτημα είναι το αν θα μπορούσαν να αναθέσουν τη διαχείριση από τα διαφορετικά ταμεία σε ιδιωτικού αισθοφορεί. Διαφορετικά δεν μπορούν να πάρουν τα κονδύλια αυτά. Ούτε καν καταλαβαίνω ποιο είναι αυτό ο ενδιάμεσο που αναφέρεται. Η ερώτηση απευθύνεται στην Επιτροπή. Το επιτρέπει ο κανονισμός. Εάν δεν εγκριθεί, πώς μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι ορισμένες χώρες δεν έχουν επαρκή ποιότητα μηχανογράφηση, συστήματο μηχανογράφηση, γιατί ξέρετε ότι η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα τα Ταμεία πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονική μορφή. Δεν στέλνουμε το, ταχυδρομείο, επί χάρτου δηλαδή τι παρατηρήσει. Ηλεκτρονική είναι η επικοινωνία. Και αν λοιπόν δεν υπάρχει το επαρκές σύστημα, αν δεν υπάρχει αντίστοιχα και υποστήριξη για τα λειτουργικά ε, προγράμματα, για τις πληρωμές, για τα μεγάλα σχέδια και για τα συστήματα ελέγχου διαχείρισης, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί ορισμένες χώρες πραγματικά δεν διαθέτουν ικανό όγκο, ε, ικανό μέγεθος για να αντιπεξέλθουν σε αυτές τις ε, τεχνολογικές απαιτήσει. Εγώ που ήμουν και από την άλλη πλευρά στο παρελθόν ως Πρωθυπουργός Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να επιτύχει κανείς για όλες τις δημοσιονομικές προοπτικές το 95%. Ο καθένα φοβόταν ότι θα τον κατηγορήσουν τα μέσα μαζική ενημέρωση ότι χάνει κονδύλιο του φεύγουν από τα χέρια, ότι δεν μπορεί να προσελκύσει τη χρηματοδότηση κτλ. Αυτό ήταν ο φόβο αποτυχία. Αλλά τώρα με τι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ μπορεί να ξεκινήσουμε μια μικρή καθυστέρηση, γιατί όταν έχουμε ένα ποσοστό μόνο 4,1% 4 δις ή από τα 200. Πολύ μικρά ποσοστά. Έχουμε φτάσει στο τέλος του 2009 και άρα πρέπει να ε, επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας. Αυτό είναι η έποψη των προϋπολογισμών. όχι ε, των, της Περιφερειακής Επιτροπής, γιατί η Περιφερειακή ε, Επιτροπή πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να επιταχύνει τους ρυθμούς της. αυτό λοιπόν που λέμε εμείς από εδώ είναι ότι τι θα κάνουμε για τα 16 δις που εκκρεμούν θα τα κατανείμουμε ή όχι, μια προοπτική. Δεύτερον, βραχυπρόθεσμα για το 2007-2013 θα μας ζητηθούν τα ποσά. Ακόμη και για το 2009 θα έχουμε αρκετά κονδύλια ή θα χρειαστούν μεταφορές. Και τρίτον, αυτές οι πραγματικές καθυστερήσεις σε ορισμένες χώρες είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν και να καταβληθούν τα κονδύλια ή όχι. Και επίσης, ναι, ξέρω, κατηγορείται πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση και η γραφειοκρατία και όλα αυτά, αλλά αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται εκεί, γιατί κάποιες χώρες μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους και κάποιε άλλε δεν μπορούν. Άρα πώ θα βελτιωθεί αυτή η πειθαρχία, αυτό ο βαθμό πειθαρχία και πώ θα αντιμετωπιστούν εκείνε οι χώρε οι οποίε τελευταία ανάλυση καθυστερούν τη διαδικασία για όλου. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τα κονδύλια και η διάθεσή του σε κάθε στάδιο τη διαδικασία. Κάποιο πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει πού πήγαν τα χρήματα και πότε. Και για ποιο λόγο. Αυτή είναι η δική μου πρόταση δηλαδή. Να ζητούμε πληροφορίε σε μηνιαία βάση να δίνονται οι απαντήσεις για το τι έχουν γίνει τα παλαιότερα κονδύλια και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την τεράστια απόκληση. Ευχαριστώ. Merci, euh, le rapporteur. Ευχαριστώ πολύ κύριε μόνιμη εισηγητά για την ε, λαμπρή και πολύ συγκεκριμένη ταυτόχρονα παρουσίαση και την ανάλυση αυτή. Η ανταλλαγή απόψεων υπενθυμίζω ότι λαμβάνει χώρα επί τη βάση μιας έκθεσης που επί προτάση του προκατόχου μου κ. Μπέγκερ ε, οδήγησε την Επιτροπή στη λήψη απόφασης για κάθε μήνα να υποβάλει έκθεση για την κατάσταση ε, ως προς την έγκριση και την εκτέλεση των συστημάτων ελέγχου διαχείρισης και των μεγάλων προγραμμάτων, των μεγάλων σχεδίων major projects των Ταμείων Συνοχής και των διαφορετικών ταμείων για το 1β δηλαδή. Γιατί διαπιστώθηκε Αφόκληση σε ορισμένα κράτη-μέλη. Πρόκειται λοιπόν για μια συζήτηση που θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε τακτικά και όπως ε, είπε και ο κύριος Κοντμάνης, πρέπει να διατυπώσουμε και τις πολιτικές, τα πολιτικά διδάγματα για τον προϋπολογισμό. Αλλά όπως προτείνει ο συνάδελφος, ίσως με, την, με το σύστημα του peer review, δηλαδή του ελέγχου από τους εταίρους, ώστε οι χώρες οι οποίες έχουν ε, καλή διαχείριση των προγραμμάτων αυτών να προσφέρουν έμπνευση με την ε, σεμνήτητα που τις χαρακτηρίζει στα άλλα ε, κράτη. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι ο κύριος Γκοντμάνης δεν αναφέρει ρητά ποια ήταν τα άλλα κράτη, οι κακοί μαθητές σε περιπτώσει. Και πρέπει εδώ, βλέποντας τα έγγραφα, να διαπιστώσουμε ότι οι κακοί μαθητές δεν είναι τα πιο νέα κράτη και ότι υπάρχουν κράτη παλαιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με γνωστή για την αποτελεσματικότητά της διοικητική δομή και γραφειοκρατική δομή, γνωστή για την αποτελεσματικότητά της υπογραμμίζω, τα οποία όμως δεν ε, είναι σε θέση να εκτελέσουν σωστά τα προγράμματά τους. Ποιος ξέρει γιατί. Θα προχωρήσω τώρα γιατί έχουμε να κάνουμε και τη συζήτηση για την πολιτική των ε, κτηρίων. Μπορούμε βέβαια κάθε μήνα να ξαναβλέπουμε το θέμα αυτό. Θέλετε το λόγο, ναι. Και τώρα παρακαλώ την κυρία Κρίσσα να το λόγο, αλλά σύντομα παρακαλώ όλοι. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Θέλω σας καλέσω στις 3.30 σήμερα το απόγευμα στην Επιτροπή Ελέγχου ε, θα έρθει ο Επίτροπος ε, για τα Περιφερειακά να μας πει για την απορρόφηση των διαστατικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού εκεί μπορούν να γίνουν και αυτές οι συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Merci Inge. Monsieur Κοτζολίνο. Κύριος Κοτζολίνο. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ δύο πραγμάτων. Τον παλιό προγραμματισμό 2000-2006 και τα αποτελέσματα αυτού του προγραμματισμού, κυρίως ως προς τις επιπτώσεις που έχουν στον προπολογισμό, το θέμα των 16 δις, ε, το οποίο επισημάνθηκε εδώ και από την έκθεση, και τη νέο, το νέο προγραμματισμό και τις επιπτώσεις που έχει ο νέος προγραμματισμός για τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι το θέμα νομίζω στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας, γνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν μας εκπλήσει το στοιχείο που μας αναφέρετε εσείς μόλις τώρα. Τα τελευταία χρόνια και μιλάω και για συγκεκριμένη εμπειρία που έχω τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία λοιπόν αυτά χρόνια ουσιαστικά ήμασταν ένα όχημα το οποίο ταυτόχρόνο έπρεπε να ολοκληρώσει το παλιό προγραμματισμό των κοινοτικών κονδυλίων ε, όπου το βασικό αίτημα ήταν να ξοδέψουμε, να επιτύχουμε ένα ποσοτικό στόχο διότι μας επέκριναν όλους για την ποσότητα των πόρων που μπορούσαμε να ε, αναλάβουμε ως υποχρέωση και να υλοποιήσουμε και ταυτόχρονα χρειάστηκε να τροποποιήσουμε το όχημα διότι οι νέοι ε, τρόποι ελέγχου μας υποχρεώνουν να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά τα ε, κονδύλια συνοχής. Και φυσικά δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό διότι όλοι οι έλεγχοι εγκρίθηκαν με ένα-ενάμιση χρόνο καθυστέρηση. Ακόμα και τις τελευταίες εβδομάδες ε, ένα μεγάλο τμήμα των κρατών μελών κατάφερε επιπλέον, ε, επιτέλους να εγκρίνει τα συστήματα ελέγχου. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, διότι περιλαμβάνει και τη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο, διότι τα κράτη-μέλη τη στιγμή στην οποία είχαμε την πιο σημαντική οικονομική και κοινωνική κρίση όπου, και όπου έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα να δαπανίσουμε με τον πιο εύκολο δυνατό τρόπο ε, τα κονδύλια, εμείς δώσαμε μια εικόνα ε, οργανωτικής μηχανής που έπρεπε να αποφασίσει πώς θα δαπανηθούν τα κονδύλια. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να προτείνω είναι να πάμε Προ την κατεύθυνση που μα υποδείχθηκε, αλλά έχοντα συνειδητοποιήσει πλήρω ότι μιλάμε για μια πολιτική ιδρυτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί την πολιτική συνοχή η Ευρώπη θα ήταν μια οντότητα την οποία θα αντιλαμβάνονταν ακόμα λιγότερο οι Ευρωπαίοι πολίτε. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ, να είμαστε ιδιαίτερω προσεκτικοί, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και μια πολιτική η οποία δεν εστιάζει τόσο πολύ στην ε, αποφυγή δεσμεύσεων, διότι αυτή ήταν μια πολιτική που ήταν κόρη της ε, ποσότητας. Αν θέλουμε λοιπόν μια πολιτική που θα ε, στοχεύει στην ποιότητα και στην καλή χρήση των κοινοτικών κονδυλίων, θα πρέπει να βλέπουμε ποια κράτη-μέλη είναι πιο καλά και να τα πρημοδοτούμε με περισσότερους πόρους και με κίνητρα που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να προχωρήσουν προς αυτή την άγουσα. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. και εσείς πραγματικά σημειώνετε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εδώ υπήρξε αλλαγή στη διαδικασία. Και αυτή η εικόνα του αυτοκινήτου, το ίδιο αυτοκίνητο που ζητάμε να κερδίσει ένα αγώνα Φόρμουλα 1 και ένα ε, ράλι παρή Ντακάρ στη Σαχάρα δεν είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Εξάλλου όλοι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα τη στιγμή της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης, όταν χρειάστηκε ε, βοήθεια, υποστήριξη η οικονομία μας, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιταχύνουμε ε, την εξέταση των σχεδίων και τη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, γιατί ήταν πάρα πολύ αυστηροί οι κανόνες μας. Και ειδού το μέγα πολιτικό παράδοξο που έχουμε ενώπιόν μας. Στον προπολογισμό του 2010 Μόλις 2,4 δις ευρώ είναι στο σχέδιο ανάκαμψης, αλλά αυτό που ε, συνεισφέρει περισσότερο στην ανάκαμψη της οικονομίας είναι όλα τα υπόλοιπα. Πολύ περισσότερο τίτλος 1β παρά η μικρή πρικοδότηση του σχεδίου ανάκαμψης. Λάσλο Σούριαν, Λαβία και μετά να περάσουμε στα κτίρια. Λάσλο. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία παρατήρηση και μία πρόταση. Is Καταρχάς είναι πολύ επικίνδυνο να πάμε στα προηγούμενα ε, για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Να σας υπενθυμίσω το non-paper. Είχαμε ένα έγγραφο το οποίο είχε πολύ ε, μεγάλες φιλοδοξίες για να πάνε εδώ, εδώ και εδώ τέλος πάντων. Πολλές από αυτές τις προτάσεις δεν θεωρούν ότι θα αυξηθεί ο προπολογισμό, θεωρούν ότι τα κονδύλια θα προέρθουν από την γεωργία ή από την πολιτική συνοχή. Και συμφωνώ απολύτω ότι χωρί την πολιτική συνοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι πλέον η ίδια. Δεν θα είναι καν Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως θα πρέπει να είμαστε φίλοι της Συνοχή. Ανεξάρτητα από το αν είμαστε από την πλευρά του δωρητή ή από την πλευρά του λαμβάνων το δώρο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε λίγο τι γίνεται. Έχουμε λιγότερο χρόνο, μας πιέζει ο χρόνος τώρα, αλλά εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμών θα πρέπει να δούμε λίγο το ρόλο μας. Ορισμένες φορές έχουμε, αν θέλετε, μία ε, οπτική από πάνω προς τα κάτω. Διαμαρτυρόμαστε, λέμε τα κράτη-μέλη δεν ξοδεύουν καλά τα χρήματά τους και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ακόμα και αυτή η μηνιαία συζήτηση μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά χρειαζόμαστε και στοιχεία. Και αυτή είναι η συγκεκριμένη μου πρόταση, μπορεί να είναι λανθασμένη, η Επιτροπή και ο Πρόεδρος ε, θα το αποφασίσει αυτό κάθε χρόνο να γίνεται μια συνεδρίαση με τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, Προπολογισμών από τα κράτη-μέλη και εκεί είναι μια ευκαιρία να ε, έρθουν αρκετές φορές. Δεν έρχεται μόνο ο πρόεδρος, μπορεί να έρθουν και οι υπόλοιποι, τα μέλη της Επιτροπής και εάν τεθεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και τους ε, ζητήσουμε αναχώρα να μας πούν για τα αποτελέσματα και τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν, τότε μπορεί να υπάρχει ε, κάποια επιρροή και για τα εθνικά κοινοβούλια. Να σας υπενθυμίσω ότι πριν από τη... μερικές ημέρες έθεσα ένα γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ρώτησα πώς εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχουμε τις πληρωμές και μάλιστα τις προκαταβολές που δίνονται. δίνουμε ένα 30% σαν δώρο και μετά από δύο χρόνια πρέπει να μας πούνε τι τα έκαναν αυτά τα χρήματα. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να μάθω πώς τα χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα, διότι σε αυτή τη φάση το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων είναι προκαταβολή. Πρόκειται λοιπόν για χρήματα τα οποία έχουν κάποιο επιτόκιο και χρησιμοποιούνται έτσι στον εθνικό προπολογισμό. Πώ έχουν τα πράγματα στην πραγματικότητα και πώ μπορούμε εμεί να ελέγξουμε γιατί χρησιμοποιούνται αυτέ οι προκαταβολέ. Για το στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, διότι η αύξηση των ε, προκαταβολών ήταν για να ε, βελτιωθούν τα πράγματα. Τώρα όμως δεν είμαστε πλέον βέβαιοι ε, εάν συμβαίνει κάτι και αν υπάρχει όντως οικονομική ανάκαμψη. Αυτή λοιπόν είναι η παρατηρήσή μου και θα ήθελα πραγματικά να συζητηθεί περαιτέρω αργότερα. Ευχαριστώ. Και μετά και εγώ δύο λόγια. Κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ όπως και ο συνάδελφος Κοτσολίνο προέρχομαι, ε, έχω την εξής εμπειρία. Έχουμε έχω συμμετάσχει σε ένα ε, πρόγραμμα ε, επιχειρησιακό για, την, ε, για τον έλεγχο των δαπανών από το 2000 έως το 2006 και θα ήθελα να επισημάνω στον εισηγητή ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα. Τα επιχειρησιακά προγράμματα των διαφόρων περιφερειών που εντάσσονται στο πρόγραμμα της πολιτικής συνοχής εγκρίθηκαν πριν από την αρχή της οικονομικής κρίσης. Και επομένως σε πολλές περιπτώσεις προβλέπουν κάποια μέτρα παρέμβασης για τους ιδιώτες οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα για τη χρηματοδότηση και τη συγχρηματοδότηση των παρεμβάσεων, που σημαίνει ότι μειώνονται οι δείκτες πρόοδου των προγραμμάτων και εδώ ε, θα ήθελα να ζητήσω και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες και να τις απλουστεύσει για τον επαναπρογραμματισμό. Διότι πολύ συχνά, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς, το πέρασμα με τη μεταφορά πόρων ε, και την ανάθεση πόρων από το ένα σημείο στο άλλο συνήθως είναι μακροπρόθεσμο και ε, φυσικά αυτό συνεισφέρει και στην καθυστέρηση των ε, δαπανών. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομα κύριε Γκοντμάνης. Ναι, δύο πράγματα μόνο. Σε σχέση με το τελευταίο σχόλιο, υπάρχει κάποιο περιθώριο. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεων από το ένα ταμείο στο άλλο. Δεν επιτρέπεται αυτό σύμφωνα με τον κανονισμό. Εάν κάποιος δεν έχει πετύχει ε, να απορροφήσει τα κονδύλια της συνοχής και θέλει να τα πάει στο κοινωνικό, δεν γίνεται αυτό. Αλλά αν η αποτυχία οφείλεται ε, στην οικονομική κρίση επειδή ένα πρόγραμμα εγκρίθηκε στο ίδιο πάντα ταμείο, μέσα έτσι στο ταμείο το διαρθρωτικό, το κοινωνικό, το συνοχής, μπορεί να γίνει μια αναδιάταξη πόρων στο εσωτερικό του ιδίου ταμείου, από το ένα έργο στο άλλο. Επαναλαμβάνω, στη συνοχή, στο κοινωνικό, αλλά όχι εγκάρσια από το ένα ταμείο στο άλλο. Βεβαίω χρειάζεται επιπλέον προσπάθεια, αλλά επιτρέπεται. Και ένα δεύτερο που θέλω να πω, ε, πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα στον προπολογισμό ως προς το εξής. Λόγω της κρίσης, τα, οι κυβερνήσεις ε, θέλουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους επιστραφούν και η διαδικασία είναι ως εξής. Όταν αρχίζει ένα πρόγραμμα, εγώ που είμαι επιχειρηματίας, ε, κερδίζω ένα διαγωνισμό. Δεν θα πάρω καθόλου χρήματα. Προκαταβολή μέχρι 4% είπε ναι ο Σούριαν, αλλά Πρέπει να πάω στην τράπεζα ή να έχω ένα κεφάλαιο και να ολοκληρώσω όλο το έργο και τότε μόνο θα πρέπει να μου πληρώσει το 75% ή ανάλογα με το ταμείο. Και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον θα έχει μαζέψει όλο το πακέτο κυβέρνηση, θα στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε και μόνο τότε θα πληρώσει την κυβέρνηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι ότι οι τράπεζε δεν είναι πρόθυμε, δεν δίνουν δάνεια και δεν έχουν αρκετά κεφάλαια οι επιχειρηματίες, είναι ταμιακό το πρόβλημα και ε, ε, ε, θέματα είναι ότι έχουν παγώσει αυτά. Δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είπε η κυρία Χιούμπνερ. Ορισμένα κράτη το διαπιστώνουν όταν αρχίζουν και τι κάνουν. Παίρνουν τα χρήματα από την χρηματοδότηση και δίνουν άμεσα δάνεια για νέα έργα. Και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, διότι συνήθως οι κυβερνήσεις πληρώνει και παίρνει την επιστροφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτει το έλλειμμά τη. Αλλά αν αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυτή την αγματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι τόνωση για να ισοσκελιστεί ο προπολογισμό, αν το δώσουν αμέσω στα δάνεια, δεν θα έχουν πρόβλημα ε, με τη χρηματοπιστωτική κρίση, θα έχουν πρόβλημα με το έλλειμμα του προπολογισμού και χώρε αρχίζουν να αλλάζουν την νομοθεσία του. Δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό δεν είναι 100% βέβαιο ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά είναι μόνο η διέξοδο, αφού δεν δίνουν λεφτά οι τράπεζε. Δεν έχουν κεφάλαια κίνηση και ταμιακή ευχέρεια οι επιχειρηματίε. Πού θα ξεκινήσει ένα έργο. Και αυτό ενδεχομένω να έχει επιπτώσει και στα δημοσιονομικά προβλήματα των κρατών πελών, μελών που επανέρχονται στον προπολογισμό τη Ένωση. Δεν ξέρω σήμερα τι... Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ. Η συζήτηση είναι πραγματικά συναρπαστική, σα διαβεβαιώ, αλλά δεν έχουμε δυστυχώ τον χρόνο να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα των κτηρίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτά. Αυτό όμω που θα ήθελα να σα προτείνω είναι το εξή. Όπως θύμισε και ο εισηγητής και οι ε, πρόκειται για τον ίδιο τον πυρήνα, την καρδιά της ε, κοινοτικής πολιτικής και τον βασικό τίτλο του προϋπολογισμού. Διότι ε, το σύνολο αυτό ε, Α και Β ε, διαρθρωτική πολιτική και ταμείο συνοχής περίπου θα καλύπτουν πλέον το 40% του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να αφιερώσουμε όλη την ικανότητα ανάλυσης και εξέταση που έχουμε. Προτείνω ο κύριος Γκοντμάνης να παραμείνει σε επαφή με τον κύριο Λαβία και τους υπολείπους που θέλουν και να προετοιμάσουν ένα σχέδιο γραπτού ερωτηματολογίου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σύνδεση με τον εισηγητή μας για τον προϋπολογισμό του 2011 και βάσει των γραπτών απαντήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πλέον να διοργανώσουμε ακρόαση με ανταλλαγή απόψεων. Όχι απλώς όπως έγινε στο παρελθόν με τους βασικούς διτρόπους ή αρμοδίους γενικούς διευθυντάς, αλλά θα πρότεινα να προσκαλήσουμε και εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, των χωρών που επιθυμούν να συμμετέχουν και είτε είναι χώρες ε, που τα πηγαίνουν πολύ καλά και έχουμε πολλά να μάθουμε από αυτές, είτε <laughs> χώρες που έχουμε να ακούσουμε πολλά από αυτές, διότι πηγαίνουν στραβά τα πράγματα για να τους κάνουμε και κάποιες συστάσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι και προτείνω να κλείσουμε εδώ τη συζήτηση και να περάσουμε στο επόμενο θέμα το 16. Ευχαριστώ την εισηγήτριά μας κυρία Χολμάγερ για την υπομονή της. Ξέρω ότι έχει εργαστεί πάρα πολύ σε δύο σχέδια πάρα πολύ διαφορετικά διαφορετικά όργανα. Πρώτον το Ίσπρα, το Κοινό Κέντρο Ερευνών στην Ίσπρα και μετά τη Βουδαπέστη. Δύο μαγικά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνικα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όντως πρόκειται για δύο μαγικά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Βέβαια είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Η πρώτη, για να το πω από την αρχή, θα το γνωρίζουν τα παλιά μέλη της Επιτροπής σε, σχέση με, σε αντίθεση με μένα, <laughs> έχουν συνηθίσει τον πόνο και τα δεινά. Εγώ αποφάσισα να μην συνηθίσω και παρακαλώ, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ περίπλοκο, παρακαλώ τη γραμματεία να έχουμε τα έγγραφα. Πρόκειται για ε, την οικοδόμηση δύο κτίριων στην Ιταλία, στην Ίσπρα για το κοινό κέντρο ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα κείμενα αυτά μόλις έφτασαν στο γραφείο μου όταν ε, ήταν σχεδόν πολύ αργά να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα για να ξέρουμε ε, όλο το ιστορικό και το υπόβαθρο. Και θα ήθελα αυτό να το απευθύνω και ρητά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι θεωρώ ότι στο μέλλον θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα και μάλιστα στο άμεσο προσεχές διάστημα. Για να αποφασίσουμε τέτοια πράγματα, μια επιτροπή προπολογισμών για να ανταποκρίνεται στα κριτήρια, να δίνει ε, βάσιμη συμφωνία, θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να γνωρίζει και το περιεχόμενο και να μπορεί να το διαμορφώνει, να έχει το χρόνο δηλαδή στη διάθεσή της, αλλιώς δεν έχει νόημα. Κατά την άποψή μου χρειάζονται αλλαγέ εδώ. Λοιπόν, έρχομαι στην ουσία. Πρόκειται για το Κοινό Κέντρο Ερευνών ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ίσπρα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη έδρα μετά τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 160 εκτάρια είναι αυτά για τα οποία πρόκειται. Τρία ε, όργανα ε, επιστημονικά 99 χρόνια από την Ιταλική κυβέρνηση το έχουμε νοικιάσει ε, προς το συμβολική τιμή του 1 ευρώ την ημέρα. Το έτος, συγγνώμη. Πριν από 5, 50 χρόνια έχουμε συμφωνήσει ε, και για την ίδρυσή του και έχουμε την 50η επέτειο. 140 κτίρια είναι και 1.800 εργαζόμενοι εκεί στο χώρο για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται και γιατί τάξη μεγέθους μιλάμε. Το 2005 ομάδα εργασίας έκανε μελέτη μετά από πενταετή αξιολόγηση στα πλαίσια του έκτου προγράμματος πλαισίου και πρότεινε ο κατακαιρματισμός των κτηρίων και ε, η δίκηση που είναι διασκορπισμένη είναι πρόβλημα και στην ε, απόδοση και στην ε, επίδοση και είναι στρατηγικό μακροπρόθεσμο το πρόγραμμα αυτό που εκπονήθηκε, ε, που μέχρι σήμερα όμως δεν είναι γνωστό σε όλους και στις λεπτομέρειές του. Θα πρέπει και εγώ να εξοικειωθώ, να το διαβάσω και ε, να ενημερωθώ. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, πρόκειται για τέσσερα νέα κτίρια που θα οικοδομηθούν για την περιβαλλοντική έρευνα, για τις επιστήμες ζωής, για την προστασία του πολίτη και την έρευνα και ένα ε, πολυλειτουργικό κέντρο συνεδρίων για να αντικαταστεθούν τα κτίρια που είναι ε, πάνω από 40 ετών για να υπάρχουν καλύτερες ε, συνθήκες όχι μόνο για τους επιστήμονες ε, στα εργαστήρια αλλά και είναι και σύγχρονα τα στάνταρ και οι προδιαγραφές ασφαλείας όπως περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό οργανισμό για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη συνεργασία των εργασομένων. Για να υπάρχει δηλαδή και θέμα χωροταξίας σε αυτό το κτίριο. Τα κτίρια που πρέπει να αντικατασταθούν τα σταθούν τώρα είναι ηλικία 40 και πλέον ετών από τη δεκαετία του 60 ε, πολύ ακριβή η συντήρησή τους και τα έξοδα λειτουργίας τους και στο παρόν θα έχουμε προσωρινές εγκαταστάσεις ε, προκάτ που χρησιμοποιούν για εργαστήρια, χωρίς να σου πω ποιος μου το είπε. Κάποιος ε, επιστήμονας μου είπε ότι έχουμε κτίρια στα οποία βρέχει μέσα και αρχίζει αυτό να γίνεται ενοχλητικό και δυσάρεστο. Επιπλέον, ορισμένα κτίρια είναι πυρηνικέ εγκαταστάσεις και στα πλαίσια ε, του προγράμματος για τον παραπλησμό τους καταστρέφονται. Εγώ γενικά ρώτησα ε, ποια είναι αυτά τα βαρύδια του παρελθόντος που μπορεί να είναι οτιδήποτε από αμίαντο μέχρι ραδιενέργεια και έχουν και χρηματικές συνέπειες. Όχι, μου είπαν τέτοια προβλήματα δεν υπάρχουν και ε, βέβαια, είμαι βέβαια ότι η τεχνολογία σε λίγα χρόνια θα μας ξεπεράσει. Λοιπόν, ε, πρόκειται για δύο κτίρια εργαστηρίων, για, εργαστήριο για τις ε, βιολογικές επιστήμες και την έρευνα για το περιβάλλον. Συνολικό εμβαδόν θα βρεθεί 27.200 τετραγωνικά μέτρα, 8.400 επιπλέον και αυτό ανταποκρίνεται μόνο στο 4%, μόλις στο 4% του συνόλου των κτηρίων της Ίσπρα. Όσο περισσότερα ε, κτίρια τώρα θα έχουμε περισσότερα εργαστήρια, ε, αίθουσες ε, συνεδριάσεων και άλλα κτίρια, άλλες εγκαταστάσεις που θα ανταποκρίνονται το καλύτερα στις σημερινές συνθήκες από τα κτίρια που υπάρχουν έγινε ένας λεγόμενος περιορισμένος διαγωνισμός, κλειστός περίπου, που ε, συμμετείχαν στην αρχή έξι επιχειρήσεις και αργότερα τρεις. Οι δύο από αυτές ήταν ε, οι πιο ε, συμφέρουσες, δεν είχαν σχεδόν καμία διαφορά και ήταν οι μειοδότες μέχρι τελευταίου λεπτού του ευρώ. Τα νέα κτίρια θα προσφέρουν χώρο για 500 άτομα διερευνήθηκε θα πρέπει να οικοδομηθούν σε μία φάση ή σε δύο φάσεις, δηλαδή ταυτόχρονα ή διαδοχικά. Η εξοικονόμηση ε, για την ταυτόχρονη ε, ε, νοικοδόμηση είναι μεγάλη και αποφασίστηκε να χτιστούν ταυτόχρονα. Τέσσερα εκατομμύρια λένε τα έγγραφά μας, δεν ισχύει αυτό ακριβώς, είναι περίπου τρία εκατομμύρια ουσιαστικά τη εξοικονόμηση. 38 εκατομμύρια είναι το κόστος και εδώ μιλούμε για το αρχιτεκτονικό, η επίβλεψη, η άδεια και 3 εκατομμύρια συν ε, μπόνους 3% για την παράδοση και 10% για την εταιρεία δηλαδή, το 3% αν παραδώσουν εγκαίρως και αυτό συμπεριλαμβάνει και τα 3 εκατομμύρια που σας είπα που ε, θα εξοικονομηθούν αν χτιστούν και τα δύο κτίρια ταυτόχρονα. Φτάνουμε λοιπόν στα 38 εκατομμύρια. 1500 ευρώ λέει κάνει το τετραγωνικό, λένε τα έγγραφα. Το συνολικό κόστος είναι 1593 για την ακρίβεια, εντάξει 1600 το τετραγωνικό. Ε, προσπαθώ να τα μεταφέρω αυτά στην πραγματικότητα. Ζητώ συγγνώμη ε, από τους συνεισηγητές μου, τους πιο συγητές, γιατί τα πήρα πολύ αργά τα στοιχεία αυτά χτες το βράδυ και δεν μπόρεσα να σας τα διαβιβάσω στο μέλλον. Θα προσπαθήσω να το αλλάξω αυτό. Τώρα, έχουμε τον εξοπλισμό τον εργαστηριακό, συν 6 εκατομμύρια περίπου δηλαδή 5.973 για την ακτήρυβια, 44 εκατομμύρια περίπου ε, το συνολικό. Λοιπόν, τώρα, ε, το σχέδιο χρηματοδότησης και εδώ αρχίζουν οι ερωτήσεις μου. Υπάρχουν έσοδα από τρίτες χώρες. Αυτά τα έσοδα από τις τρίτες χώρες ετησίως ανέρχονται σε 12 εκατομμύρια ευρώ. Πρόεδρος Διακόπτη, συγγνώμη κυρία εισηγήτρια, διότι Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Κατανοώ ότι για το πρόβλημα της ίσπρα έχουμε χρόνο. Θυμίζω στους συναδέλφους, ζητώ Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ, λέει η κυρία Χολμάγερ. Λοιπόν, θυμίζω στους συναδέλφους ότι πρόκειται για το άρθρο 179.3 του κανονισμού, του δημοσιονομικού κανονισμού. Κάθε φορά λοιπόν που ένα οποιοδήποτε θεσμικό όργανο έχει ένα κτηριακό ε, σχέδιο ενημερωνόμαστε και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι αν θέλουμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα και να γνωμοδοτήσουμε. Και έχουμε 15 μέρες για να πούμε ναι ή όχι. Εντάξει. Αν ναι, έχουμε επιπλέον 15 μέρες. Συν Χριστούγεννα και γιορτές και διακοπές για να γνωμοδοτήσουμε. Εξ όσων έχω καταλάβει, ε, κυρία Συγκητρία, για την Ίσπρα έχετε ακόμα ερωτήσεις να υποβάλλετε και θα προτείνετε στην Επιτροπή Προπολογισμών όντως να εφαρμόσουμε το άρθρο και να κάνουμε γνωμοδότηση. Αυτή είναι η πρότασή σας. Αυτό θα προτείνετε. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε, γιατί ήθελα απλώς να σας εξηγήσω πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα και γι' αυτό κατά την άποψή μου θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Ιανουάριο να βάλουμε την απόφασή μας γιατί και το θέμα των διαγωνισμών και της χρηματοδότησης χρειάζεται να το ξαναδούμε. Άκουσα ότι οι συνεισηγητές, οι σκιώδες ηγητές ε, έχουν την ίδια άποψη και θα ήθελα να αναβολή ακριβώς για να ε, μπορέσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Ζήτησε εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, όχι, ζήτησαν δύο συνάδελφοι, ο κύριο Βόγκαν και ο κύριο Μάνκα, το λόγο να μιλήσουν. Προτείνω να ακούσουμε του συναδέλφου αυτού και ενδεχομένω και άλλου, που να κάνουν όμω ερωτήσει ή σχόλια, αλλά να έρθετε αμέσως σε επαφή με την κυρία Χολμάγερ μετά τη συνεδρίασή μας. Να βεβαιωθώ ότι η Επιτροπή Προπολογισμού συμφωνεί να ασχοληθούμε με το πρόβλημα και να γνωμοδοτήσουμε. Να συνεχίσουμε δηλαδή τη συζήτηση και να την ολοκληρώσουμε με ψηφοφορία στην επόμενη συνεδρίαση. Και στο μεταξύ όλοι οι συνάδελφοι που θα είχαν ερωτήσει να κάνουν, να κάνουν προτάσεις να ενημερωθούν. για να έχουμε ακριβώ χρόνο τώρα για να ασχοληθούμε με το άλλο πρόβλημα που πρέπει σήμερα να αποφασίσουμε, νομίζω, που είναι η εξαγορά του κτηρίου στη Βουδαπέστη. Ε, συμφωνείτε? Ωραία. Ποιο συμφωνεί λοιπόν να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή μας για την Ίσπρα, να ασχοληθεί με το θέμα λοιπόν, αλλά για τον Ιανουάριο. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Υποθέτω Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Χολμάγερ και σα ζητώ συγγνώμη που επιταχύνω λίγο τα πράγματα, αλλά όπω καταλαβαίνετε έχουμε ε, τώρα ε, την υποχρέωση και παρουσία του αρμοδίου αντιπροέδρου στο προέδρου ε, του κύριου Βιντάλ Κουάδρα να ασχοληθούμε με ένα σχέδιο που είναι κατεπήγον και μάλιστα σε πολύ προχωρημένο στάδιο η εξαγορά του κτηρίου στη Βουδαπέστη για το Κοινοβούλιο. Η κυρία Χολμάγερ. Κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι προβληματικό, είναι λιγότερο προβληματικό. Χαίρομαι που ήρθε ειδικά ο πρόεδρος για να το συζητήσουμε και να μας ενημερώσει πώς έχει κατάσταση. Εγώ θα είμαι σύντομη. Πρόκειται για το έτος 2008 η προϊστορία. Για ποιο λόγο φτάνει με τέτοια επίγουσα ε, πλέον ε, πίεση, γιατί έπρεπε να έρθει τον Ιανουάριο αυτό το θέμα είναι ότι προσπαθούμε να το βάλουμε στο προπολογισμό του 2009 ακόμα και είναι η τελευταία συνεδρίαση για να έχουμε περιθώριο λιγμό στο προπολογισμό του 2010. Γι' αυτό μπήκε τόσο απότομα και τόσο νωρί στην ημερήσια διάταξη και πρέπει να αποφασιστεί κιόλα. Πρόκειται για το εξή θέμα. Στη Βουδαπέστη τώρα εμεί τι θέλουμε θέλουμε να έχουμε αλλαγή στρατηγικής. Δηλαδή, μέχρι τώρα τα γραφεία ενημέρωσης ήταν πάντα γραφεία που αγόραζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμμετείχε ε, κατά 40%. Τώρα αλλάγει η στρατηγική, το ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέγει δεν μπορεί να αγοράσει το Κοινοβούλιο το κτίριο και να μας πληρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 60% έχετε μια καλή περιγραφή των κτίριων στους φακέλους σας. Πρώτον έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια και επίσης το κτίριο είναι πιο αντιπροσωπικό, ε, προσωπευτικό ε, σε κεντρικό σημείο και με μεγάλη προβολή. Και θα ήταν ε, προνόμιο αυτό και πλεονέκτημα και για τον Ουγγρική Προεδρία. 130 ευρώ κοστίζει σήμερα το τετραγωνικό για έξοδα και στο νέο είναι 70 ε, ευρώ το τετραγωνικό και μεγάλη εξοικονόμηση. Έχουμε και χαμηλότερο κόστος ενέργειας και ε, έχουν και όλα τα κτίρια επιτέλους και όλα τα γραφεία φυσικό φως ε, παράθυρα. Και Θα γίνει μειοδοτικό ε, διαγωνισμός για τη διαχείριση σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Κανονισμό. Χρηματοδότηση θα έρθει από το αποθεματικό για τα κτίρια του 2009, άρθρο, ε, ε, τίτλος 5, ε, συγγνώμη, κεφάλαιο 105 και σήμερα θα πρέπει να αποφασίσουμε. Προϋπολογίζεται 10,1 εκατομμύρια, εκατομμύρια το κτίριο, 7,19 είναι το αντίτιμο και όλα τα άλλα είναι τα έργα που χρειάζονται. 100.000 υπάρχει περιθώριο και ένα εκατομμύριο για να πληρωθεί ε, το κόστος ε, των ε, δικηγόρων και βασικοί φόροι μάλλον ε, για να εγγραφεί στο υποθηκοφυλακείο κτλ. Ευχαριστώ κύριε Σίτρη. Ο κύριος Χάγκλουντ θέλει το λόγο και ο αντιπρόεδρος θα μας πει την άποψή του. Πολύ σύντομα για τη διαδικασία. Εχθές το βράδυ είχα επιτέλους τη δυνατότητα εξ ονόματος της ομάδας μου να εξετάσω λίγο την υπόθεση της Βουδαπέστης. Μου φαίνονται καλά τα πράγματα. Το μόνο που θα ήθελα να πω σε αυτή τη φάση είναι ότι όπως είπε και η κυρία Χολφμαϊερ πριν, ως νέο μέλος μου φαίνεται λίγο περίεργο να δεχτώ το γεγονός ότι όταν μιλάμε για ακίνητα λαμβάνουμε όλες τις πληροφορίες στην τελευταία στιγμή. Και επειδή είμαι και σκιώδης συγητής για την πολιτική ακινήτων, δεν ήταν τόσο εύκολο να τα εξετάσω, γιατί έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Και όταν λαμβάνετε όλη την, ε, ε, την ύλη για αυτά τα, τα κτίρια την προηγούμενη μέρα, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά μας. Θα ήθελα απλώς να τα λαμβάνω λίγο νωρίτερα, ώστε να έχω και τη δυνατότητα να έχω μια πιο σαφή εικόνα γιατί αποφασίζουμε. Ήθελα να το πω και ελπίζω να μην συμβαίνει το ίδιο για όλες τις περιπτώσεις ακινήτων, γιατί και για την κυρία Χολμάγερη, αλλά και για μας θα είναι πολύ δύσκολη η δουλειά μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, για το κτίριο τα πράγματα είναι καλά και χαίρομαι που και οι Ούγγροι συνάδελφοι είχαν τη δυνατότητα να το δουν το κτίριο και τους ικανοποιεί. Ε, ελπίζω λοιπόν να προχωρήσουμε, αλλά ελπίζω στο μέλλον να μας δίνονται πληροφορίες ε, νωρίτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γιατί θα έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω όταν ξεκινήσει η διαδικασία, όταν τεθεί σε ισχύ. Αλλά ήταν πολύ εύστοχη η παρατήρηση. Ο κύριο Μάνκα όμω έχει στήσει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ με την συγκεκριά αλλά και με τον προλαλήσαντα. Εδώ και πέντε χρόνια βλέπουμε ότι έρχεται τελευταία στιγμή μια πληθώρα πληροφοριών. Δεν είναι σοβαρό τρόπο αυτό να επεξεργόμαστε την κατάσταση, την κατάσταση και γι' αυτό θα ήθελα να δω πώ θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δεν είναι σοβαρό αυτό ο τρόπο. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν. Το καλύτερο θα ήταν να κάνουμε αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί, κάθε δηλαδή ε, θεσμικό όργανο να προσδιορίζει τη δική του μέσο και μακροπροθέσμια προοπτική, στρατηγική να γίνεται ο συντονισμό και να γίνεται σε τελικό, στο τελευταίο στάδιο ο τελικό συντονισμό μεταξύ όλων των ε, θεσμικών οργάνων. Έχω μια ερώτηση όμως να πόσο Το Κοινοβούλιο, από ό,τι φαίνεται, ήθελε να αγοράσει το κτίριο και μετά η Επιτροπή σκόπευε να καταβάλει τα ποσά στο Κοινοβούλιο. Κάπως ανετράπη δηλαδή η διαδικασία. Πώς έγινε αυτό. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Αντιπρόεδρος θα ήθελε παρακαλώ να λάβει το λόγο, να μας εξηγήσει τις ε, παρατηρήσεις στα σχόλια. Να δώσει απαντήσεις πριν προχωρήσουμε στην απόφαση. Ah, yes. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η κυρία Νομίζω ότι η κυρία Ολπαγέρ εξήγησε αρκετά καλά το σχέδιο. Πλην όμως, για αυτή τη φορά ακολουθούμε μια μέθοδο κάπως ασυνήθιστη. Αγοράζουμε δηλαδή εμείς και μας αποζημιώνει η Επιτροπή το 60%. Συνήθως γίνεται το αντίστροφο. Αγοράζει η Επιτροπή και εμείς αποζημιώνουμε κατά 60%. Συμμετέχουμε κατά 60%. Ερώτηση χωρίς μικρόφωνο. Για λόγους συγκεκριμένους η Επιτροπή είχε δυσκολία αυτή, τη στιγμή, αυτή την εποχή να, κάνει την, ε, να προβεί στη συναλλαγή αυτή. Μας ζήτησε λοιπόν να προβούμε εμείς στην αγορά και μετά θα μας επιστρέψει αυτό το ποσοστό, το 60% επί το μου του χρόνου. Δεν θα νοικιάσει, θα καταβάλει το 60% επί το μου. Καλώς. Άρα η κατάσταση από ό,τι φαίνεται είναι λίγο παράδοξη του χρόνου, του χρόνου, του χρόνου. Το ταχύτερο δυνατόν. Είναι κάπω ε, ιδιαίτερη κατάσταση. Ο κύριο Βιδάλ Κουάντρας μέχρι 31 Δεκεμβρίου έχει λεφτά. 31 Δεκεμβρίου τέρμα τα χρήματα. Άρα, εάν δεν πάρουμε την απόφασή μας αμέσω, χάνουμε τα, τα λεφτά αυτά. Από την άλλη, η Επιτροπή το 2009 δεν έχει λεφτά, αλλά θα έχει από την 1η Ιανουαρίου του 2010. Μα εξήγησε ο κ. Βιδάλ με ένα πολύ ωραίο τρόπο υποβίβαση, αν θέλετε, τη σοβαρότητα κατάσταση, μάλλον καταλανική έμπνευση, ότι βρισκόμαστε σε μια παροδική αδυναμία ε, ρευστότητος. Αυτό που προτείνει λοιπόν η Σύγητρια είναι να μην θέσουμε σε λειτουργία το άρθρο 169, δηλαδή να γνωμοδοτήσουμε θετικά. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Δίνουμε το πράσινο φως με το να μην γνωμοδοτήσουμε δηλαδή. Πλην όμως μόνο και εδώ στρέφονται όλα τα βλέμματα με θαυμασμό και προσδοκία στον κύριο και τον άνθρωπο κλειδί που ήρθε με υπομονή και άντεξε τόσες ώρες και τον ευχαριστούμε για την απαντοχή του, που όμως τώρα και εδώ ενδυναμώνεται ο, η ανησυχία και η, αδυνομία, και η δημονία, να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Κύριε Λεβαντόφσκι, προφανώς, προφανώς έχει λογική αυτή η λύση γιατί χρήματα έχουμε, μπορούμε να απορροφήσουμε το αποθεματικό για τα κτίρια και να το ενισχύσουμε του χρόνου με 6 εκατομμύρια όταν θα έχουν ε, ληφθεί αποφάσεις για τις προσαρμογές στη Λισαβόνα. Δημοσιονομικά βεβαίως είναι λογική αυτή η λύση. Δεδομένου ότι εκπνέει μίσθωση στην Βουδαπέστη και ακολουθεί άλλωστε και η Ουγγρική ε, προεδρία, άρα όλα νομίζω συγκλίνουν υπέρ αυτής της μεταφοράς. αριθμών 24 όμως. Mm. Ναι. C'est un mariage, je l'aime, elle... Ωραία. Δηλαδή, ε, ευτυχία με, αυτή την, με αυτό τον ιερό δεσμό με αγαπάει, την αγαπώ, συμφωνούν και οι γονείς και ως εκ τούτου το 2009 αναλαμβάνει το βάρος του Κοινοβούλου, το 2010 η Επιτροπή. Καλώς 24 υπέρ, ευχαριστώ, κατά ουδείς αποχές. Ζήτω! Αγαπητοί συναδελφοί, σας ευχαριστώ. Και αφού εξαντλήσαμε την ανεξάρτητη μερίσια μας διάταξη, σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Χάρη δε στην ποιότητα των εισηγητών και των συζητήσεων έγινε μια συναρπαστική ανταλλαγή απόψεων και όπως είπα και νωρίτερα, μάλλον αντίθετα από ό,τι είπα αρχικά προβλέποντας ε, τις εξελίξεις, καταλαβαίναμε τι ψηφίζαμε. Προσεχή συνεδρίαση δεν γνωρίζω πότε θέλω να Γιατί προβλέπετε με την ακρόαση του υποψηφίου Επιτρόπου επί θεμάτων προπολογισμού για τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Οπότε θα προβλεφθεί έκτακτη συνεδρίαση. Έχουμε όμως υπόψη ότι η τακτική συνεδρίαση προβλέπεται για την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ πολύ και πέρα στις συνεδριάσεις